So, since the in the room, Μια και είναι εδώ η για Γιάνν Όλμπριχτ, ας ξεκινήσουμε. So, meine Damen und και κύριοι, Καλώς ήρθατε στην απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ο κύριος Σαρτουή, πρόεδρος, σας ενημέρωσε το πρωί ότι δεν θα μπορούσε να παραστεί και έτσι έχω εγώ τη χαρά να τον αντικαταστήσω στην Προεδρία της Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη το οποίο θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο Πρόκειται για την ευελιξία στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και εδώ καλωσορίζω την κυρία Εουλάλια Ρούμπιο και τον κύριο Πέτερ Μπέκερ. Χαίρομαι που είστε εδώ. Για να μας προσφέρετε τη φώτα σας στα θέματα αυτά. Έχουμε δύο γραπτές τοποθετήσεις, ενημερωτικά έγγραφα από πλευρά σας. Θα δώσω το λόγο και στο Richard Κρότ της Νομικής Υπηρεσίας που έχει εκπονήσει για το θέμα αυτό μελέτη. Και ρωτώ τον κύριο Ολμπρίχτ, αν θέλετε εσείς κύριο Ολμπρίχτ να λάβετε πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ. Ε. Σήμερα εκπροσωπώ και την κυρία Τωμάτη, συνεισηγήτρια. Και θα κάνω μία σύντομη εισαγωγή για το που βρισκόμαστε. Ε, εκπονούμε την έκθεση πρωτοβουλίας ε, που θα υποβληθεί το Φεβρουάριο στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στο έγγραφο αυτό Θα εξετάσουμε πρώτα κάποια βασικά στοιχεία από την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενδιάμεση αξιολόγηση. Πρώτον. Δεύτερον, από το ψήφισμά μας για το μελλοντικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα έχουμε κάποια στοιχεία και επίσης ε, θα λάβουμε και κάποιες προτάσεις από τις κοινοβουλευτικέ επιτροπές που ε, εκπονούν τις δικές τους γνωμοδοτήσεις για το ΠΔΛΤΑΠΗ. Στο δικό μας, στη δική μας έκθεση θα κάνουμε πρώτα κάποιες γενικές παρατηρήσεις για το χαρακτήρα του προϋπολογισμού, τη δομή του προϋπολογισμού, φυσικά και τη διάρκεια του, αλλά και κάποια στοιχεία που αφορούν το όλο οικοδόμημα και την αρχή της ευελιξίας ή κάποια στοιχεία της ευελιξίας. Θα ασχοληθούμε λοιπόν και με την ευελιξία και με την ενότητα του προϋπολογισμού. Γιατί από την αρχή ήδη προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την ευελιξία του προπολογισμού, καθιστώντας τον πιο ανοιχτό και πιο εύπλαστο κατά την επταετία αυτή. Γι' αυτό ένα από τα στοιχεία που προτείνουμε είναι ε, τι είδου ε, μηχανισμούς έχουμε που ήδη λειτουργούν εύρυθμα και συνάδουν με την ευελιξία και ποιοι τέτοιοι μηχανισμοί θα πρέπει να διορθωθούν, να ανανεωθούν, ενδεχομένως θα χρειαστούμε και κάποιους νέους μηχανισμούς ευελιξίας ή κάποια νέα στοιχεία ευελιξίας. Οπότε θα δούμε τι λειτουργεί από την ε, ισχύουσα ευελιξία και τι μπορεί να αλλάξει ή να βελτιωθεί. Επίση, η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προ την ενότητα του προπολογισμού. Όταν μιλούμε για την ενότητα του προπολογισμού, φυσικά η Επιτροπή μα, η Επιτροπή Προπολογισμών, ανακάλυψε στο μέτρο που προχωρούσε την περιπλοκότητα τη χρηματοοικονομικής δομής και δεν θα έλεγα μόνο τη δημοσιονομική δομή, γιατί ναι μεν μιλούμε για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Υπάρχουν και κάποια ε, συμπαρομαρτούντα θέματα. Οπότε υπάρχει ένα ολόκληρο στερέωμα στοιχείων αλληλένδετων γύρω από τον προϋπολογισμό και με τον προϋπολογισμό. Οπότε θέλουμε να διαμορφώσουμε μια καθαρή εικόνα. Α, αυτό που έχουμε στον προπολογισμό να αντικατοπτρίζει τις πολιτικές, γιατί θα πρέπει να δούμε τι πολιτικές θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε από κοινού τι εργαλεία, τι μηχανισμούς έχουμε και να εξετάσουμε κατά πόσο ο προπολογισμό αντικατοπτρίζει το πλέγμα, το, τη δέσμη πολιτικών που η συνθήκη αποφάσισε να ε, χαραχθούν από κοινού. Επίσης, θέλουμε να δούμε τον πραγματικό ρόλο των εξωτερικών ε, μηχανισμών και να εξετάσουμε, να εξακριβώσουμε κατά πόσο χρειαζόμαστε τέτοιους εξωτερικούς μηχανισμούς. Μήπως μπορούμε κάποια χρηματοοικονομικά κάποιου κάποιους χρηματοοικονομικούς εξωτερικού μηχανισμού θα του συμπεριλάβουμε στον προπολογισμό. και ποιε θα είναι οι συνέπειε, γιατί πολλέ φορέ λέμε αν περιλάβουμε κάτι τέτοιο στον προπολογισμό, χωρί να αλλάξουμε τα ανώτατα όρια, κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει τον προπολογισμό. Οπότε ε, θα πρέπει να διαρωτηθούμε αν τα χρειαζόμαστε, αν χρειαζόμαστε τέτοιους μηχανισμούς, αν ε, καθιστούν το σύστημα πιο ευέλικτο, αν διανοίγουν νέε δυνατότητε, ή μήπω είναι απλώ ένα επιπλέον στοιχείο χωρί όμω πραγματική προστιθέμενη αξία γιατί έτσι προσθέτουμε μια σειρά στοιχείων και στο τέλος χάνουμε τον έλεγχο σε αυτά. Επίσης, διαρωτόμαστε για το ρόλο των μηχανισμών αυτών και τη σημασία τους. Και επίσης, κατά πόσο ελέγχουμε αυτού του μηχανισμού. Εμεί είμαστε ερετό σώμα, μπορούμε να ελέγξουμε ή θα έπρεπε να ελέγξουμε αυτούς τους μηχανισμούς. Μήπως ε, τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να ε, υπάρχει τέτοιο κοινοβουλευτικό έλεγχο σε τέτοιου μηχανισμού. Και αυτά όλα τα πραγματευόμαστε και αυτά τα δύο στοιχεία αποτελούν το αντικείμενο και τη σημερινή ακρόση. Πρώτον, ευελιξία στο πλαίσιο του νέου πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου και δεύτερον, το θέμα τη ενότητα του προπολογισμού. Και ελπίζουμε με την ακρόαση αυτή να συγκεντρώσουμε όχι μόνο πληροφορίες αλλά και προτάσεις και συστάσεις για να τις συμπεριλάβουμε στο εγγραφό μας. Ευχαριστώ κύριε Ολμπρίχτ. Έχετε λοιπόν κυρία Ρούμπιο πολλές ερωτήσεις και από τον εισηγητή και από την Επιτροπή μας. Περιμένουμε ενδιαφέρον να ακούσουμε τις προτάσεις σας ελπίζοντας ότι θα μας δώσετε και απαντήσεις. Έχετε το λόγο. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω, θα σας παρουσιάσω ένα σύντομο σημείωμα για, την, για το επόμενο ΠΔΕΛΤΑΠΗ και την ευελιξία. Να κάνω μια επισκόπηση της παρουσίασης. Καταρχήν θα σας ε, δώσω μια ε, γενική προσέγγιση των σκέψεών μας για, την, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα παρουσιάσω κάποια τις διατάξεις ε, περί ευελιξίας. Ε, θα εξετάσουμε κατά πόσο οι ισχύουσε διατάξει ευελιξία λειτουργούν στο παρόν ΠΔΠ και κάποια θέματα για τη χρήση της ευελιξίας στο πλαίσιο 2014-2020 και κάποιου τρόπους για να διευρυνθεί, η, ενισχυθεί η ευελιξία στο επόμενο ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ μετά το 2020. Καταρχήν να σας δώσω τη δική μου εντύπωση για το ποιες θα είναι οι βασικές προκλήσεις του επόμενου ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ. Θα μπορούσαμε ε, να συνοψίσουμε τις προκλήσεις σε μια διπλή πρόκληση. Καταρχήν θα πρέπει να προσαρμοστούμε στο μόνιμο χρηματοδοτικό κενό που θα αφήσει το Brexit, γιατί με την ε, αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα δημιουργηθεί μια ένα κενό που έχει υπολογιστεί γύρω στα 10 δισεκατομμύρια το χρόνο γιατί αποχωρεί ένας ε, αμυγής συνεισφορέας και θα έχουμε αυξημένες δαπάνες λόγω νέων προτεραιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια, μετανάστευση. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων δεν είναι εύκολη. Το πιο εύκολο ή το πιο επιθυμητό σενάριο είναι να βρεθούν νέοι πόροι για να γεμίσει αυτό το κενό, να γεφυρωθεί με νέου ενδεχομένω πόρου ή νέου ίδιου πόρου, διαφυλάσσοντα το ισχύον επίπεδο ε, πληρωμών ή να έχουμε μια μετάβαση ε, ή μεταφορά πιστώσεων προς ε, νέες πολιτικές από τις παλιές πολιτικές και ο καλύτερος τρόπος να το κάνουμε θα ήταν με έξυπνες και εκβάθρο μεταρρυθμίσεις στις δύο τομείς πολιτικής, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και μειώνοντας τις συνολικές δαπάνες. Ιδιαίτερα στις δύο πολιτικές συνοχής και γεωργική. Είναι το επιθυμητό σενάριο, αλλά πολύ αμφιβάλλω θα μπορούσα να το υλοποιήσουμε μέχρι το 2019. Οπότε ένα εναλλακτικό σενάριο θα ήταν ένα μεταβατικό πι με κάποιες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να μειωθούν οι προϋπολογισμοί στη συνοχή και την ε, ΚΑΠ. Ε, βέβαια, οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε δύο βασικούς τομείς πολιτικής ενόψη και των επόμενων ευρωεκλογών θα είναι κάπως δύσκολο εγχείρημα γιατί λίγος χρόνος υπάρχει ε, και θα πρέπει να ετοιμαστούμε ε, για το επόμενο ΠΔΠ. Οπότε το δεύτερο πιθανό σενάριο είναι κάποιες μεταρρυθμίσεις και μεταβίβαση πόρων από, τις από τις παλιές τις νέες ε, πολιτικές και ε, να ξεκινήσουμε μια πιο ρηξικέλευτη μεταρρύθμιση του σύστηματος ιδίων πόρων αν μη τι άλλο να εγκριθεί μέχρι το 2019. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παρούσα ευελιξία και τις ε, διατάξεις περί ευελιξίας και πώς χρησιμοποιούνται στο ισχύον ΠΔΠ. Υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις από αυτήν την άποψη. Καταρχήν προτάθηκαν ε, διατάξεις ε, ευελιξίας για να μεγιστοποιηθεί η χρήση των περιθωρίων πληρωμών αναλήψης υποχρεώσεων και του περιθωρίου απρόβλεπτων αναγκών και κάποια εγγενής ευελιξία ε, στο αποθεματικό έκτακτης ανάγκης, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύη, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής ε, στην Παγκοσμιοποίηση και επίσης έχουμε τέτοια γενή ευελιξία σε κάποια προγράμματα δαπανών. Τώρα, πώς ε, τα ειδικά, ειδικοί μηχανισμοί βρίσκονται στο ΠΙΔΑΛΤΑΠΗ Καταρχήν, διαπιστώσαμε ότι έχουμε εκτενή χρήση του μηχανισμού ευελιξίας, που ήταν ο μηχανισμός που κατεξοχήν ε, χρησιμοποιήθηκε και ήταν και ο πιο ενδιαφέρον και εύκολος να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Χρησιμοποιήθηκε το 2015 και το 2016 με αποτέλεσμα το 2016 να έχουμε εξαντλήσει το διαθέσιμο ποσό του μηχανισμού ευελιξίας, ενώ στους άλλους μηχανισμούς έγινε πιο μετριοπαθής και άνηση αξιοποίηση και χρήση τους. Κάτι άλλο που μπορούμε να λάβουμε υπόψη είναι ότι ο κανονισμός του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ δεν ήταν σαφής ό,τι αφορά τη μεταχείριση των δαπανών για τη χρήση των μηχανισμών αυτών. Κάτι που προκάλεσε συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπιστούν, πώς θα χειριστούμε αυτές τις ε, πληρωμές. Θα πρέπει να είναι εντός των ανώτατων ορίων ή να εξαιρούνται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις θεώρησε εκτός των ανώτατων ορίων. Κατά τη γνώμη ήταν θετική αυτή η απόφαση, γιατί αν τις πληρωμές αυτών των μηχανισμών τις εντάξουμε στα ανώτατα όρια, κάθε φορά που κινητοποιούμε τους μηχανισμούς αυτούς, μειώνουμε ακόμη περισσότερο τα διαθέσιμα περιθώρια για τις επόμενες χρονιές. Οπότε καλώ δεν τα περιέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα περιόρισε πολύ την ευελιξία. Έχουμε και κάποιου πίνακε για τη χρήση των ειδικών αυτών μηχανισμών, αλλά θα τους ε, περάσω. Αν σας ενδιαφέρει μπορείτε να τους κοιτάξετε στις διαφάνειες που τις τυπώσαμε και όλα και να θέσετε σχετικές ερωτήσεις, γιατί για την παρουσίαση δεν έχω πολλή ώρα. Περνάμε τώρα στις ε, διατάξεις ευελιξίας για τη μεγιστοποίηση της χρήσης των περιθωρίων. Αυτή ήταν και η βασική καινοτομία του ΠΔΠ. Το περιθώριο πρόβλεπτων αναγκών επέτρεπε την αύξηση των ε, των πιστώσεων πληρωμών και ανάληψη υποχρεώσεων με βάση το ΑΕ ε, και επίσης μειώνεται τη χρησιμοποίηση ε, ε, του ολικού περιθωρίου για υποχρεώσεις και για πληρωμές και η δυνατότητα μετάβασης στα επόμενα χρόνια και χρήση των δύο περιθωρίων. Τώρα, μπορούμε να συνάγουμε κάποια συμπεράσματα. Καταρχήν, τα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν από το ολικό περιθώριο για τις υποχρεώσεις και για τις πληρωμές ήταν ε, πολύ μεταβλητά αυτά τα ποσά από το ένα χρόνο στο άλλο, ανάλογα με το περιθώριο. Σε μερικές χρονιές είχαμε σημαντικά περιθώρια και σε άλλες όχι τόσο. Σε ό,τι αφορά το περιθώριο απρόβλεπτης ανάγκης, ε, απρόβλεπτων αναγκών που σχετίζεται με το ακαθάριστο ε, χώριο εισόδημα είναι πιο προβλέψιμο. Βέβαια, η χρήση του περιθωρίου απρόβλεπτων αναγκών θα πρέπει να αντισταθμιστεί από πόρους των επόμενων χωρών. Οπότε, γίνει εκτενής χρήση του περιθωρίου απρόβλεπτων αναγκών για μία χρονιά, περιορίζονται τα περιθώρια από υποχρεώσεις και πληρωμές στις επόμενες χρονιές θα έχουν περιοριστεί πολύ τα περιθώρια, τα ολικά περιθώρια υποχρεώσεων και πληρωμών για τις επόμενες χρονιές. Οπότε θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια διόρθωση στη συνέχεια μετά την αύξηση αρχικά. Τώρα δούμε την... το γενικό περιθώριο για τις υποχρεώσεις, για τις πληρωμές, συγγνώμη, είναι μια καινοτομία και εξασφαλίζει μέγιστη χρήση των συνολικών, πληροφοριών, των συνολικών πληρωμών. Και αν δείτε τη γραφική αυτή παράσταση βλέπετε δύο στοιχεία. Την πάνω γραμμή είναι το τρέχον πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και η κάτω γραμμή είναι η προηγούμενη περίοδος 2007-2013. Η γαλάζια γραμμή είναι οι πιστώσεις πληρωμών που εγκρίθηκαν τη στιγμή της θέσπισης του ΠΔΠ και η κόκκινη γραμμή είναι οι πιστώσεις πληρωμών με βάση την τελευταία τεχνική προσαρμογή. Και κάτω έχετε το ίδιο τις συγκεκριμένε πιστώσεις πληρωμών σε μπλε κατά τη στιγμή της θέσπισης του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ και στη κόκκινη γραμμή τις πληρωμές την τελευταία χρονιά του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ Βλέπετε πολλές αναξιοποιητά κονδύλια που δεν χρησιμοποιήθηκαν και άρα επιστράφηκαν στα κράτη-μέλη. Και τώρα, στο ισχύον ΠΔΕΛΤΑΠΗ δεν θα έχουμε κάτι τέτοιο, γιατί όταν είχαμε μείωση των πιστώσεων από το 2016 δεν μπορούν να ανακτηθούν αυτές οι αναξιοποιητές ε, δαπάνες. Γιατί συνήθως τις τελευταίες χρονιές του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ έχουμε αύξηση των απαιτήσεων. Άρα πρέπει να βελτιστοποιηθεί το συνολικό περιθώριο για τις πληρωμές. Σε ό,τι αφορά το ολικό περιθώριο για τις υποχρεώσεις, αυτό δεν έχει δώσει και πολύ σημαντικά ποσά. Ήταν χρήσιμο, αλλά θεωρούμε ότι το γενικό περιθώριο για τις υποχρεώσεις περισσότερο χρησιμοποιήθηκε για να ανταποκριθεί στην ευελιξία που οφειλόταν στο γεγονός ότι το ΠΔΠ δεν συγχρονιζόταν με τη διάρκεια των, της θητείας και του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό και δημιουργήθηκαν νέε προτεραιότητε, χρειάστηκαν και νέα κονδύλια. Οπότε το ολικό περιθώριο για τι υποχρεώσει δεν χρησιμοποιήθηκε παρά για να ε, χρηματοδοτηθεί μία αλλαγή, μία καμπή στις πολιτικές προτεραιότητες. Σε ό,τι αφορά την εγγενή ευελιξία των προγραμμάτων δαπανών, ε, είχαμε σταδιακές προσαρμογές σε κονδύλια της συνοχής, ε, βέβαια είναι σχετικά άκαμπτη αυτή η δαπάνη γιατί το 70% των δαπανών έχουν προσημειωθεί αλλά υπάρχει μια εγγενής τέτοια ευελιξία σε κάποια προγράμματα πληρωμών, δαπανών μάλλον. Τώρα, ποια είναι τα σημαντικότερα μαθήματα κατά τη χρήση των και εφαρμογή των διατάξεων της ευελιξίας. Διαπιστώνουμε ότι η ευελιξία εξαρτάται από την ύπαρξη επαρκών περιθωρίων. Αν έχουμε διατάξεις ευελιξίας που συνίστανται στη χρήση περιθωρίων κυρίω, τότε θα πρέπει να έχουμε επαρκή περιθώρια για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτέ τι διατάξει. Και αν δείτε τι γίνεται στι διαπραγματεύσει του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ, έγινε μια συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου. Γιατί ε, το Συμβούλιο ήθελε χαμηλά όρια και για πληρωμέ και για υποχρεώσει. και τελικά ενώ ήταν αρχικά αρνητικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δέχτηκε σε αντάλλαγμα κάποιες διατάξεις ευελιξίας. Τελικά δεν ήταν και πολύ καλή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η συμφωνία αυτή, γιατί η ύπαρξη περιθωρίων είναι προϋπόθεση για την ευελιξία. Χωρίς περιθώρια, όσο ωραίες και αν είναι οι διατάξεις περί ευελιξίας, είναι άχρηστες εφόσον δεν υπάρχουν περιθώρια. Γιατί, επαναλαμβάνω, η ευελιξία στηρίζεται σε περιθώρια, οπότε χωρίς περιθώρια δεν υπάρχει ευελιξία. Επίσης, το θέμα της μεταχείρισης των πληρωμών που απορρέουν από τη χρήση ειδικών μηχανισμών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποίησε μια πιο ευνοϊκή ερμηνεία προ τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά καλό θα ήταν στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο αυτό να διευκρινιστεί. Και επίση το θέμα τη ενδιάμεση αξιολόγηση. Ε, βέβαια, έγινε συζήτηση ε, και έγινε η παρουσίαση για το επόμενο ΠΔΠ. Αν θα έχουμε ένα ΠΔΠ μεγαλύτερη διάρκεια, θα πρέπει σε τέτοια περίπτωση η ενδιάμεση αξιολόγηση να είναι ουσιαστική και να δημιουργήσει δυνατότητα για τις απαραίτητες αλλαγές. Κάτι που δεν συνέβη στην δική μας περίπτωση λόγω των ε, νομικών περιορισμών. Δεν μπορούσαμε να τροποποιήσουμε ε, τα ανώτατα όρια ή προσημειωμένα κονδύλια. Τώρα πώς θα ενισχύσουμε την ευελιξία. Στο έγγραφο ε, εξετάζω κάποιες προτάσεις για παράδειγμα, με κάποιες αλλαγέ στη δομή και τη διάρκεια του ΠΔΠ. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε γιατί ε, αυτό δεν αφορά ε, μόνο τη διαρθρωτική και ε, τη διάρθρωση και τη διάρκεια. Πάντως για ευελιξία, όταν έχουμε μικρότερο αριθμό τομέων, η δυσκολία μεταβίβασης κονδυλίων από το ένα τομέα στον άλλο θα είναι πιο δύσκολη. Τώρα, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τους ειδικού μηχανισμούς εκτός του ΠΙΔΑΛΤΑΠΗ. Ε, είδαμε ότι είναι οι μηχανισμοί ευελιξίας χρήσιμοι και θα μπορούσαμε να δούμε αν μπορούμε να συγχωνεύσουμε μερικούς μηχανισμούς. Για παράδειγμα, ε, να συγχωνεύσουμε το μηχανισμό ευελιξίας με το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας. Επίσης, προτάθηκε η σύσταση ενός αποθεματικού κρίσης. Είναι μια πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη στην ενδιάμεση αξιολόγηση. Βέβαια, ένα αποθεματικό έκτακτης βοήθειας μπορεί να καλύψει κάπως ή να συμπληρώσει ένα αποθεματικό κρίσης, οπότε θα είχε νόημα μια τέτοια συγχώνευση. Ένας άλλος τρόπος ενίσχυσης είναι με τους περιορισμούς ό,τι αφορά τη μεταβίβαση κονδυλίων από τη μια χρονιά στην άλλη. Μέχρι στιγμής μπορεί να γίνει μεταφορά ε, ενός τμήματος των ανα, μη χρησιμοποιημένων κονδυλίων. Δεν ξέρω βέβαια αν θέλουμε κάποιους κανόνες αποδέσμευσης ε, για τη, τις πολιτικές δαπάνες. Για μηχανισμούς πάντως που η κινητοποίησή τους εξαρτάται από το κατά πόσο συμβαίνει όχι ένα προσδόκητο γεγονός, δεν ξέρω αν έχει νόημα να, να περιορίζουμε τη δυνατότητα χρήσης αναξιοποίητων κονδύλιων. Γιατί επειδή μια χρονιά δεν χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο αυτό, δεν, δεν βλέπω γιατί να μας περιορίζει τις επόμενες χρονιές που ίσως έχουμε περισσότερες ανάγκες. Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στις ε, υφιστάμενες διατάξεις ευελιξίας, όπως είπα, η προϋπόθεση για το ρόλο, σημαντικό ρόλο των διατάξεων ευελιξίας είναι η ύπαρξη επαρκών περιθωρίων. Βέβαια, μπορούμε να ενισχύσουμε τις διατάξεις αυτές. Σε περίπτωση του περιθωρίου των αναγκών θα μπορούσαμε ε, να καταργήσουμε τη δυνατότητα αντιστάθμισης ε, των κονδυλίων που χρησιμοποιήθηκαν από τις επόμενες χρονιές. Οπότε ανακτούνται όλα τα ποσά που είχαν περιλαμβάνοντα τη διοργανική συμφωνία πριν τη συνθήκη της Λισαβόνα και που δίνουν τη δυνατότητα τροποποίηση του ΠΔΠ μέχρι ενό βαθμού, μέχρι 0,003% με το Συμβούλιο να λαμβάνει απόφαση με ενισχυμένη πλειοψηφία. Οπότε θα είχαμε μια πιο ευκίνητη διαδικασία του, της τροποποίησης του ΠΔΠ για μικρά σχετικά ποσά. Μία πιο καινούργια πρόταση εδώ είναι η πρόταση της δημιουργίας ενός δημοσιονομικού αποθεματικού σε κάθε ε, κοινοτικό προϋπολογισμό. Οπότε όλοι οι αιτήσιοι προϋπολογισμοί πάγονται σε υποχρεωτικά ε, περιθώρια. 5% ε, ε, των δαπανών που δεν χρησιμοποιηθεί να μπαίνει στον ετήσιο προϋπολογισμό και έτσι να δημιουργηθεί ένα αποθεματικό με, αυτές τις, με αυτά τα χρησιμοποίητα ποσά και για να κινητοποιηθεί το αποθεματικό αυτό θα πρέπει να λαμβάνουν απόφαση οι αρμόδιες για τον προπολογισμό αρχές. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί ένα αποθεματικό μία χρονιά θα μπορούσε το ποσό του να τροφοδοτήσει το ολικό περιθώριο για τις υποχρεώσεις ή το γενικό περιθώριο για τις πληρωμές. θα μπορούσαμε εύκολα να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο δημοσιονομικό αποθεματικό. Το αρνητικό σημείο είναι ότι περιορίζει τα ποσά για τα προγράμματα. Οπότε χρειαζόμαστε επαρκή ανώτατα όρια για να επιτραπεί η χρήση τέτοιων υποχρεωτικών περιθώριων. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ähm, ευχαριστώ κυρία Ρούμπιο. Κύριε Ούλριχ, θέλετε εσείς το λόγο. Ο συγητής λαμβάνετε πρώτος το λόγο. Ιδάλλως ο κύριος Ρούμπιχ και ο κύριος Φερνάντες που μου έχει στείλει το λόγο. Κύριε Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε λεπτομερώς τις ε, δυνατότητες εναλλακτικέ που έχουμε. Νομίζω ότι η σημειοκίνηση πρέπει να είναι πάντα η συνθήκη της Λισαβόνας. 1,24% προβλέπει, άρα πρέπει να γίνει συζήτηση ε, η θεμελιώδη συζήτηση πώς θα εξασφαλιστεί η υλοποίηση του 1,24% επί του ΑΕΠ που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Και πάλι. Και πώς μπορούμε να τηρήσουμε αυτό το οποίο έχει ήδη συμφωνηθεί. Αυτή είναι η ουσία. Πρέπει να δούμε ποια προγράμματα είναι σημαντικά. Για παραδείγματι, εγώ στην Επιτροπή μου έχω ιδιαίτερα το θέμα της ε, ε, αναπτυξιακής πολιτικής και εκεί μπορούμε να πούμε σε ποιους διακυβερνητικούς τομείς ε, μπορούμε να επεκτείνουμε τον ε, τακτικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ποιοι είναι οι διακυβερνητικοί εκείνοι τομείς και διεθνή ακόμη προγράμματα που μπορούν να συμπεριληφθούν στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη οι διαπραγματεύσεις από το Brexit θα ορίσουν κάποια συγκεκριμένα ποσά. Ένα συγκεκριμένο ποσό, ανεξαρτήτως του ύψους του, που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει ότι πρόκειται για ένα δις ευρώ, ότι πρέπει να πάρουμε ένα δις ευρώ ε, με την ολοκλήρωση του Brexit, ιδάλλως δεν πρόκειται να εγκρίνουμε το Brexit. Είναι μια σκληρή γραμμή για μας βέβαια και πρέπει να ξέρουμε αν δεν τα καταφέρουμε τι δυνατότητες αναδίπλωσης έχουμε. Ε, και επίσης αυτά τα 100 δις θα πρέπει σταδιακά, λίγο-λίγο, τμηματικά να ξαναμπούν μέσα στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Με ποιους όρους θα γίνει αυτό. Το αναπτυξιακό ταμείο, το Brexit, αλλά και πολλοί άλλοι τομείς πρέπει νομίζω να διευκρινιστεί πώς θα ε, εκτελεστούν μέσα από τις προϋποθέσεις του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με νέες ανάγκες, όχι μόνο με το ε, αναπτυξιακό πρόγραμμα υπαριθμών νέα αλλά και με την γεωργία και με, τις, ε, με τη διαφορετική πολιτική. Άρα τίθεται πάντα το ερώτημα αυτής της ευελιξίας. Αυτή πρέπει να θέσουμε στο επίκεντρο των συζητήσεών μας και έχουμε τη δυνατότητα και για το μέλλον μαζί με το Συμβούλιο να αναπτύξουμε μια θεώρηση για το μέλλον. Ο κύριος Μακρόν της Γαλλίας ε, έχει ε, εντάξει ως ύψιστη προτεραιότητα το θέμα αυτό στο πρόγραμμά του και καλό θα ήταν να μην συνεχίσουμε ως Ευρώπη τις παλαιές και γνωστές παραδόσεις κάθε χρόνο να μειώνουμε λίγο, να ε, συστέλουμε λίγο τον προϋπολογισμό ώστε να φτάσει να είναι και κάτω από το 1% επί του ΑΕΠ ε, για να εκτελέσει, να επιτελέσει τα σημαντικά του καθήκοντα. Εάν θέλουμε στο μέλλον αυτά τα σημαντικά καθήκοντα να τα επιτελεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός πρέπει να εξασφαλίσουμε και τις δυνατότητες για να το πράξει αυτό. Και πάντα υπάρχουν κάποια τμήματα στη διοίκηση που υπολογίζουν πόσα δισεκατομμύρια χάνουμε ε, χρήματα του Ευρωπαίου πολίτη, επειδή δεν κάνουμε από κοινού κάποιες πράξεις, από κοινού, και χτυπώ την κροθιά στο τραπέζι, από κοινού κάποιες δράσεις, αν θέλουμε μια Ευρώπη ισχυρή, πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να αποδείξουμε αποτελεσματικότητα με όλη την επικουρικότητα βεβαίως, αλλά υπάρχει μεγάλο κόστος από την απουσία της Ευρώπης, από το non-Europe. Και αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Η συνθήκη της Λισαβόνας έχει βεβαίως αναπτυξιακή πολιτική, γεωργία, διαρθρωτική πολιτική. Αυτές είναι οι βασικές της προτεραιότητες. Δεν μπορούμε να υπολοιπόμεθα των αναγκών και πρέπει στον κύριο Μπαρνιέ με απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο να πείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να δεχθεί Brexit εάν δεν εξασφαλιστούν τα 100 ε, Ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για το κείμενο, ευχαριστώ τη μελέτη, την παρουσίαση για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που είναι η ευελιξία. Είναι κάτι που οι διαπραγματευτές αγωνίστηκαν γι' αυτό και κέρδισαν. Και είναι πολύ σημαντικό και για το Συμβούλιο και την Επιτροπή ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως αυτά που είχαμε με τους πρόσφυγες. Και είναι απίστευτο πόσο δυσκολευτήκαμε. Για το θέμα τώρα του επιθυμητού σεναρίου. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν είναι επιθυμητό όμως και το οποίο μάλιστα αντιβαίνει και στην εσωτερική αλληλεγγύη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ε, υπάρχει μια πολιτική, δύο μάλλον, που λειτουργούν καλά, είναι εκείνη της συνοχής και η... εκείνη της κοινή γεωργικής πολιτικής. Το να τις μειώσουμε μπορούμε, όλα μπορούμε να τα μειώσουμε. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν αυτή η σωστή προσέγγιση. Και πολλές φορές τα βάζουμε με την πολιτική συνοχής, ενώ γνωρίζουμε ότι σε αυτό το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο φέτος το 2017 ουσιαστικά αρχίζει για το 2014, 2015 και 2016 είχαμε ε, να πληρώσουμε από το προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και θα συνεχίσουμε και το 2021, 22 και 23 επίσης, γιατί έχουμε τον κανόνα νη συν 3. Αν λοιπόν κοιτάξουμε από το 2017 μέχρι το 2023, θα δούμε ότι θα υπάρξει μια εξαιρετική χρήση του προπολογισμού. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το 1,23 νομίζω που είναι το ανώτατο ή 1,24 για τις πληρωμές. Πρέπει όμως να πούμε 1,23 το ανώτατο δηλαδή που αποφασίστηκε για ίδιους πόρους σε πληρωμές, ναι, σε πληρωμές γιατί είναι ένα 27 σε υποχρεώσεις, έτσι. Λοιπόν, αναρωτιέμαι αν αυτό είναι η σωστή προσέγγιση και μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε αν αυτό πρέπει να είναι το ποσό που πρέπει να έχουμε για τον προπολογισμό. Υπάρχουν προφανή ζητήματα. Αλλά ας δούμε πού πάμε τελικά. Να μειώσουμε την περίοδο, να βάλουμε ένα χρόνο. Θα μπορούσαμε. Όχι εμείς, εντάξει, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο υπάρχει το άρθρο 312 της συνθήκης της Λισαβόνας που λέει ότι το ελάχιστο είναι πέντε χρόνια. Αλλά λέω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι για να έχουμε την ανώτατη ευελιξία μπορούμε να βάλουμε ένα χρόνο. Γιατί σε πέντε χρόνια πάλι δεν μπορούμε να προβλέψουμε πράγματα ούτε για μετά από ένα-δύο χρόνια. Είναι αυτά τα πρόβλεπτα που λέμε. Άλλοι λένε να μειώσουμε τον αριθμό των τομέων. Να βάλουμε έναν και να τα βάλουμε όλα μέσα. Ορίστε. Μέγιστη ευελιξία αυτή. Έτσι δεν χρειάζεται προβλεψιμότητα για τις περιφέρειες, δεν χρειάζεται προβλεψιμότητα για τους δικαιούχους. Και γι' αυτό τα εθνικά κυρίως κονδύλια και τα κονδύλια για τα προγράμματα είναι σημαντικά. Αλλά υπάρχει μια ιδέα που μου αρέσει. Να πούμε να αλλάξουμε το όνομα να μην το λέμε ότι είναι περιθώριο για τα πρόβλεπτα και να το κατανέμουμε σε επόμενες χρονιές. Οπότε δεν θα αφαιρούμε ένα πρόβλεπτο, θα ξεκινάμε από την αρχή που λέει ότι πρέπει να χρηματοδοτείτε από νέο χρήμα. Για τελειώς κόβουμε τις άλλες προτεραιότητες αν έχουμε ένα πρόβλεπτο. Είναι μια καλή ιδέα και αυτή που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, να εξετάσουμε. Και κάτι ακόμα για τα δημοσιονομικά ε, μέσα. Για το Συμβούλιο οι πληρωμές είναι μέσα στον προπολογισμό. Για την Επιτροπή τα ειδικά μέσα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εκτός προϋπολογισμού. Όλοι γνωρίζουν ότι αν έχουμε υποχρεώσεις εκτός προϋπολογισμού, αυτό σημαίνει ότι και οι πληρωμές είναι εκτός προϋπολογισμού. Για το Συμβούλιο, που του αρέσει πάντα να τα κόβει όλα, τους αρέσει να λένε όχι, είναι μέσα στον προϋπολογισμό. Ακόμα και αν είναι πεπισμένοι ότι είναι εκτός προϋπολογισμού. Ευελιξία λοιπόν, πολύ σημαντικό θέμα. Και δεν ξέρω μήπως η καλή λύση είναι να πούμε χρειαζόμαστε περιθώρια, αφήνουμε μεγάλα περιθώρια για να έχουμε ευελιξία. Τότε το Συμβούλιο πάντα θα έχει τάση, και όχι μόνο το Συμβούλιο, να λέει δεν θα πειράξουμε το περιθώριο αυτό για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για την ευελιξία. Αλλά υπάρχει μια αρχή που έχει λειτουργήσει καλά και είναι το συνολικό περιθώριο για τις υποχρεώσεις, για τις πιστώσεις υποχρεώσεων και αυτό πρέπει να το έχουμε. Και να έχουμε και άλλη μια αρχή που λέει ότι κάθε ευρώ το οποίο προβλέπεται στον προπολογισμό πρέπει να παραμένει στον προπολογισμό. Στις πιστώσεις υποχρεώσεων και στις πιστώσεις πληρωμών. Και υπάρχει και κάτι που πιστεύω ότι δεν είναι σοβαρό, είναι σε πληρωμές να έχουμε ένα ποσό το οποίο να είναι κατά πολλά δισεκατομμύρια χαμηλότερο από το ποσό που έχουμε στις υποχρεώσεις. Γιατί αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος, το Συμβούλιο, που πάντα ελπίζει ότι δεν θα χρειαστούμε αυτό το χρήμα. Υπάρχει αυτή η ευτυχής ιδέα ότι εμείς δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα. Αλλά αυτό θα πρέπει να απαλληφθεί ως ιδέα ότι προβλέπετε, να προβλέπετε με την ιδέα ότι κάθε ευρώ στον προπολογισμό που εγγράφεται θα πρέπει και να χρησιμοποιείτε. Και σε υποχρώσεις και σε πληρωμές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκόλμ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά παρακολούθησα την παρουσίαση της κυρίας Ρούμπιο και πρέπει να πω ότι κάποια σημεία με ενοχλούν τώρα κάποιες παρατηρήσεις. Φερρυπίν, κύριε αν μου επιτρέπετε να απευθύνω σε εσάς το λόγο. Λέτε ότι πρέπει να πληρώσουν 100 ε, εκατομμύρια ευρώ οι Βρετανοί για τον Brexit. Ε, έχω μήνες τώρα ζητάω να μου δείξει κάποιος μια μέθοδο υπολογισμού. Έχετε κάποια μέθοδο εσείς ή απλώς είπατε σας αρέσει το ποσό που είναι στρογγυλό και λέτε 100 δις. Ας είμαστε λίγο σοβαροί όμως. Θέλω να δω με ποιον τρόπο υπολογισμού καταλήγεται στα 100 δις. Γιατί εάν όντως έχουμε λογαριασμούς εκρεμής ανοιχτούς για 100 δις, έχω την εξής ερώτηση. Και να είμαστε πάλι γενναιόδοροι και να στρογγυλοποιούμε τα ποσά, οι Βρετανοί συμβάλλουν με, με 10% στον προπολογισμό μας. Το υπόλοιπο 90% το καλύπτουν οι υπόλοιποι. Φεύγουν τώρα οι Βρετανοί και έχουν 100 δις χρέος, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι έχουν 900 δις χρέος συνολικά. Ε, άλλα 9 δις, 3 ε, μάλλον χρέος, πού τα βρήκατε. Ας μην κάνουμε κουβέντες του αέρα τώρα, ε, ας κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση και να ζητούμε όντως τα χρήματα τα οποία οφείλουν οι Βρετανοί. Και επίσης ε, ομολογώ ότι όντως είναι αλλεργικές οι αντιδράσεις μου. Καμιά φορά όταν ακούω κάτι δηλώσει ότι χρειαζόμαστε τώρα ποσά. Σαν να ε, ισχύει το ρητό ότι ό,τι είναι ακριβό είναι και καλό. Ε, όχι, νομίζω ότι πια πρέπει να κοιτάξουμε να καταρτίζουμε έναν προπολογισμό ο οποίο να στοχεύει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και αυτό με την επεξεργασία του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου πρέπει να είναι ο στόχος μας, να ορίσουμε πρώτα απ' όλα καλούς στόχους, αλλά καλή στόχη είναι αυτοί οι οποίοι είναι και μετρήσιμοι. Δεν αρκεί δηλαδή να πούμε «Α, περιγράφω κάτι ωραίο, μου φαίνεται καλό, συμφωνώ και το περιγράφω έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορώ να θεωρώ ότι εκτελώ και το στόχο». Όχι, πρέπει να είναι σαφή οι στόχη. Γιατί λοιπόν, εξηγήστε μου, η γεωργική και η πολιτική, ε, η διαρθρωτική, σε ποιο βαθμό ικανοποιούν τους στόχους μας. Χρήμα μοιράζουμε με τη γεωργική πολιτική. Αυτό είναι ο κύριος στόχος όλης της ε, επιχείρησης και στην ε, πολιτική συνοχής. Έχουμε πολύ καλά μέτρα, αλλά έχουμε και άλλα μέτρα τα οποία επί δεκαετίες δεν επιτελούν το στόχο τους. Εάν λοιπόν επί δεκαετίες δεν έχουν φτάσει στο στόχο τους, είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι όλα είναι καλά, δεν πρέπει να το αμφισβητήσουμε. Και γι' αυτό τώρα με την επεξεργασία του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, πρέπει να κοιτάξουμε αυτή τη διάσταση. Ευχαριστώ κύριο Μπούγκερ. Ε, ευχαριστώ. Όλα φαίνονται τόσο εύκολα και απλά. Είναι απλό όμω το πράγμα. Το, η υπόθεση του Brexit είναι απλή. Μπορούμε να κάνουμε από κοινό τον υπολογισμό. Να πούμε συμφωνούμε αυτό που χρειάζεται. Ένα ε, απλό ετήσιο προπολογισμό και το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο στο, έως το 2020 για τι υποχρεώσει και έως το 2023 για τι πληρωμέ. Και ο κύριο Ρουμπίχ πολύ σωστά επισημαίνει ότι καθαρό εισφορέ του προπολογισμό όπω το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μια αμφίροπη σχέση με τον ε, προϋπολογισμό. Έχουμε την έκπτωση της εκπτώσεως, ένα άλλο θέμα, πολύ επίκυρο αλλά όντως είναι ο, κατά έτος κατά 11 δισεκατομμύρια εισφορέας στον προϋπολογισμό. Ας δούμε τώρα τα μεγάλα αυτά κεφάλαια που αναφέρατε κι εσείς. Γεωργία, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ε, Γεωργική Ανάπτυξη, Ανάπτυξη της Υπέθρου. 700 δις ευρώ για την διάρκεια ολόκληρη, δηλαδή ένα 100 ε, δις ανά έτος. Απλός υπολογισμός. Βγάζω δέκα που είναι το δύσκολο. Δεν καταραίει ο ευρωπαϊκός προπολογισμό με το Brexit. Ούτε και εξάνισταται τα πνεύματα για το τι είδους ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα πρέπει να έχουμε μετά το Brexit. Νομίζω ότι υπάρχει επαρκής επιστημονικός τρόπος υπολογισμού που να λέει τόσο δίνεις κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό, φεύγεις τώρα και άρα με αυτή την μέθοδο υπολογισμού φτάνουμε μεταξύ των 60 και των 100 δις, γιατί είναι και οι συντάξει μέσα. Αλλά σε όλη αυτή τη συζήτηση ένα πράγμα δεν ε, αναφέρεται και δει στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναφέρεται ότι το ζήτημα δεν είναι μια κίνηση ανθρωπισμού. Είναι μια κίνηση που έχει να κάνει με το σεβασμό στις δεσμεύσεις, στις διεθνείς συνθήκες, τη Διεθνή Σύμβαση της Βιέννης για τις Διεθνείς Συμβάσεις. Για κοιτάξτε τα σχετικά άρθρα, γιατί αναφέρεται ξεκάθαρα ότι είναι ε, υποχρεωμένος όποιος αποχωρεί από μια διεθνή συνθήκη ή σύμβαση να τηρεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Και όσο είναι μέσα είναι υποχρεωμένος και να τηρεί αυτά τα οποία έχει αναλάβει ως δέσμευση. Άπαξ και αποχωρήσει δεν δεσμεύεται πλέον. Για να σας το πω αλλιώς, όποιος φύγει από το κοπάδι χωρίς να έχει εκτελέσει το, το καθήκον του, με βάση το διεθνές δίκαιο, είναι δυνατόν να είναι ένας ε, συνομιλητής με τον οποίο θα έχω εμπιστοσύνη να συνάψω νέα σύμβαση, νέα συνθήκη. Και ένα άλλο, κάπως πιο νεφελώδες πεδίο, γιατί έχουμε να κάνουμε με τις διεθνείς joint ventures, την Ίσπρε παραδείγματι, όπου υπάρχει κοινή χρηματοδότηση με διεθνούς δικαίου δεσμεύσεις πλέον. Τι τις κάνω εγώ αυτές τις joint ventures. Τον Γαλιλαίο. Τι το κάνουμε. Πώς υπολογίζουμε το γεγονός ότι είναι νομική προσωπικότητα, ότι έχει νομική προσωπικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου έχει δικαίωμα στην ιδιοκτησία και έχει την ιδιοκτησία ενός δορυφόρου και θέλουν οι Βρετανοί να συνεχίσουν να έχουν μέρος, ε, να λαμβάνουν μέρος σε αυτό το έργο. Και αν κάποιο δορυφόρο δεν δουλεύει, τι κάνουμε. Λοιπόν, είτε συμμετέχουν σε κάποια συγκεκριμένα σχέδια με το σύστημα που έχουμε για την Νορβηγία, είτε αποχωρούν. Η Νορβηγία κάθε χρόνο πληρώνει 900 εκατομμύρια ευρώ, υποστηρίζοντας τα ασθενέστερα κράτη συνοχής στο, στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό η Νορβηγία και αντίστοιχα συμμετέχει σε 4-5 προγράμματα στα οποία έχει μέρος. Έχει λάβει μέρος. Άρα, εάν θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσει να συμμετέχει και στην καινοτομία και την έρευνα, με τα 10 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίω που επωφελούνται των ερευνητικών, από τα 10 μάλλον καλύτερα παγκοσμίω, τα τρία είναι βρετανικά, επωφελούνται από το, από το Ταμείο Έρευνα και Καινοτομία. Αν είναι έτσι, συνεχίζει να πληρώνει, ιδάλω χαίρεται. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε και να δούμε από εκεί και πέρα τις περαιτέρω συμφωνίες, νέες συμφωνίες που θα είναι και πιο δύσκολο να γίνει ο υπολογισμός γιατί θα πρέπει να προσδοριστεί και η μελλοντική σχέση συνεργασίας. Αλλά αυτά που ισχύουν μέχρι τώρα είναι ξεκάθαρα και σαφώς υπολογίσιμα. Και αυτό σας λέω και πάλι ότι δεν σημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός Προπολογισμό, σε περίπτωση hard Brexit καταραίει επειδή δεν συμφωνήσαμε με τους Βρετανούς. Αλλά έχω και κάποιες ερωτήσεις κυρία Ρούμπιο για τις πρώτες αναλύσεις ε, και τα επιθυμητά σενάρια για μεγάλες μεταρρυθμίσει στο τομείο Συνοχής, στη γεωργική πολιτική. Και ναι και ου. Διότι συγκρούσεις μεταξύ των ε, κεντρικών των, ε, των μεγάλων αστικών κέντρων, ε, των μητροπολιτικών κέντρων της, του, του κάθε κράτους μέλους με την περιφέρειά τους και την ύπεθρό τους μπορεί να ενισχυθούν σημαντικά εάν αυτά όλα καταρριφθούν. Πώς λοιπόν θα λειτουργήσουμε, πώς θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αυτή τη ζημιά με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ανοίγουμε δηλαδή νέα πεδία σύγκρουσης και βρισκόμαστε ενώπιον του μεγάλου προβλήματος της βιωσιμότητας και τη απασχόληση και τη ανάπτυξη και των άλλων των μεγάλων ε, έργων μα. Λοιπόν, βεβαίω να κοιτάξουμε πού μπορούμε να κάνουμε οικονομία, πού μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πώ απορροφούνται από ορισμένα κράτη τα κονδύλια, πώ μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική η περιγραφή και πιο συγκεκριμένη ω προ τι διαστάσει του των προγραμμάτων και των έργων που αναλαμβάνουν κάποια κράτη, να είναι πιο καλά προσαρμοσμένα στι ανάγκε του και τι δυνατότητε του με τι συστάσει. Ναι, μέχρι εκεί καλά. Και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διπλασιάζουμε, τριπλασιάζουμε τον ευρωπαϊκό Προπολογισμό, Όπως είπε και ο Πάουλ Ρουμπίχη, έχουμε ε, επίπεδα. Έχουμε ανώτατα επίπεδα, το δημοσιονομικό πλαίσιο αφενός και τους ίδιου πόρους αφετέρους. αφετέρου. Και αυτά ούτω ή άλλω θα υπάρχουν, σύντο χρόνο θα τα έχουμε πάντα. Από εκεί και πέρα, το περιθώριο το οποίο κανεί δεν συζητάει χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο βρίσκεται σε αμηχανία, δεν ξέρει τι πρέπει να κάνουμε από εκεί πέρα, δεν έχει τρόπο χρηματοδότηση. Κοιτάει να δει αν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις, τις εγγυήσεις της ε, ΕΤΕΠ, του μέσου υποστήριξης κτλ. Εκεί που δεν υπάρχουν τα 50-60 δις που μας χρειάζονται. Τρία κράτη εκτός του ευρώ έχουν, της Ευρωζώνης έχουν σε περίπτωση κρίσης αξιοποιήσει τέτοια κονδύλια και αν λοιπόν έχουμε συγκεκριμένες προκλήσεις για την μακροπροθεσμή σταθεροποίηση της εξωτερικής πολιτικής, της διασφάλισης των συνόρων, όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν με το εφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρέπει να εξηγήσουμε στα κράτη-μέλη γιατί το ζήτημα της ασφάλειας είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει τα κράτη-μέλη να εξηγήσουν γιατί είναι ένα ζήτημα αυτό της ασφάλειας που είναι διατεθειμένα να αμφισβητήσουν. Και πρέπει να το εξηγήσουν στους πολίτες. Και επίσης Έχουμε προσπαθήσει μερικές φορές αλλά δεν καταφέραμε ποτέ τα κράτη-μέλη να ανοίξουν έναν δρόμο και να πούν ότι φτιάχνουμε ευρωπαϊκούς οργανισμούς ή ε, συνάπτουμε ευρωπαϊκά έργα ταυτόχρονα με αναδιάρθρωση των εθνικών δομών. Με αμφισβήτηση ακόμα και του γεγονότος ότι μπορεί να μην χρειάζεται ένα Εθνικό Υπουργείο, εάν υπάρχουν οι άλλες δομές. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να τα κοιτάξουμε και να τα πούμε στους εθνικούς δημοσίους υπαλλήλου και τις γραφειοκρατικές δομές των κρατών μελών. Επίσης ε, υπήρξε ζήτημα ε, σε σχέση με την ε, με την ανακατανομή 2015-2016 που κινδύνευσε το πολιτές νομικό πλαίσιο το τρέχον να καταρρεύσει. Αυτό πρέπει να είναι ένα μάθημα και πρέπει να κοιτάξουμε να αναζητήσουμε και άλλες δυνατότητες διεύρυνσης της ευελιξίας, να τις μελετήσουμε προσεκτικά και να είμαστε έτοιμοι γνωρίζοντας τι θα φέρει η κάθε εξέλιξη και να μην χρειάζεται κάθε φορά σε περίοδο κρίσης να περνάει ένας μήνας ή και περισσότεροι για να καταλήξουμε κάπου. Τώρα λοιπόν αυτή η μεταρρύθμιση πρέπει να είναι μια πραγματική, μια πραγματική αναθεώρηση με την πραγματική έννοια της λέξης και να κοιτάξουμε με βάση το δημοσιονομικό δίκαιο και τα όσα ορίζει οπωσδήποτε η συνθήκη της Λισαβόνας τι έχουμε χάσει σε σχέση με αυτά και να τα μελετήσουμε πολύ προσεκτικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ. Εξαντλήσαμε έτσι τον κατάλογο των ομιλητών. Κύριε Λέναρτ, δεν ε, σας καλούμε να δώσετε απαντήσεις για κάθε ζήτημα που αφορά τις δημοσιονομικές μας σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, για το πόσο βαθιά θα βάλουν το χέρι στην τσέπη, αλλά μιλήστε μας λίγο για την ευελιξία και τοποθετηθείτε, αν θέλετε βέβαια, στα όσα μας είπε η κυρία Ρούμπιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. θα μπορούσα να σχολιάσω τα περί υποχρεώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Όσον αφορά όμως την ευελιξία, η εντύπωσή μου είναι από τις διάφορες συζητήσεις ότι υπάρχει μια ασυνήθιστη συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για το ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να δούμε αν μπορούμε να την ενισχύσουμε περισσότερο αυτή την ευελιξία. Θα συμφωνούσα με αυτά που τόνισε ο κύριος Ρουμπίχ και που είπατε ότι έχουμε διανύσει πολύ δρόμο και η επιπλέον ευελιξία, ας είμαστε ειλικρινείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να την πετύχει στον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων και είναι πολύτιμη αυτή η επιτυχία και για τις υποχρεώσεις και για το περιθώριο απρόβλεπτων. Πράγματι, πού θα ήμασταν σήμερα αν δεν είχαμε αυτές τις καινοτομίες στην εφαρμογή. Πάντα βέβαια ακολουθώντα και τη λογική που λέει ότι αν δεν μπορούμε να έχουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα θέλαμε, τουλάχιστον να χρησιμοποιήσουμε μέχρι το τελευταίο σεντ το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που καταφέραμε να έχουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορούμε βέβαια να σκεφτούμε και άλλες βελτιώσεις παρετέρω την επόμενη φορά, την μεθεπόμενη και για τα ειδικά εργαλεία και για το ότι πληρωμές πρέπει να είναι πάνω από την οροφή και η Επιτροπή θα προτείνει σαφές κείμενα από αυτού. Είναι η μόνη λογική προσέγγιση αυτή. Όσον αφορά τώρα τα περιθώρια, θέλω να ρωτήσω και, τον κύριο, και την κυρία Ρούμπιο και άλλους να κάνουν ε, μια διάκριση στα περιθώρια στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και στον ετήσιο προπολογισμό. Τα περιθώρια στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πολύτιμα γιατί με τα νέα μέσα, τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, δημιουργούμε και πάλι την ετήσια διαδικασία προπολογισμού η ετήσια δημοσιονομική διαδικασία έχει περιοριστεί στο χρόνο, ακριβώς επειδή υπάρχει πολλής ε, προπρογραμματισμός ε, του προπολογισμού. Ενώ τώρα με τα περιθώρια μπορούμε κάθε χρόνο να δουλέψουμε πάνω σε αυτά. Αυτά για τα περιθώρια στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στον ετήσιο προπολογισμό όμως, ο προπολογισμό πρέπει να χρησιμοποιείται και ό,τι είναι διαθέσιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Εντάξει, θα μπορούσαμε να αφήσουμε λίγο περιθώρια για την επόμενη χρονιά, αλλά είναι δύσκολο να κινητοποιηθεί με τροποποιητικές διαδικασίες. Οπότε είναι πολύτιμα τα περιθώρια στο πολιτικο δημοσιονομικό πλαίσιο, όμως το ετήσιο προπολογισμό όχι γιατί οι δυνατότητες δαπάνησής τους είναι ελάχιστες. Επίσης θέλω να επιστήσω την προσοχή στο ρόλο του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου ως συνομοθέτες. Έχετε εσείς τη δυνατότητα να ορίσετε την ευελιξία μέσα σε προγράμματα κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Και τα προγράμματα τα οποία εγκρίθηκαν την προηγούμενη φορά σε μερικές περιπτώσεις έχουν προβλέψει μέχρι 100% τη χρήση των κονδυλίων. Ας πούμε για το παράδειγμα γειτονίας, τα κονδύλια επανακατανεμήθηκαν στις δικιούχους χώρες 100%. Αυτό βέβαια δεν βοηθάει δεδομένου ότι οι προτεραιότητες μιας περίοδου αλλάζουν. Η εξωτερική πολιτική κατάσταση αλλάζει. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να πείσει τους νομοθέτες την επόμενη φορά να αφήσουν κάποια περιθώρια και μέσα στα προγράμματα ώστε να μπορούν να αντιδράσουν αν χρειαστεί σε απρόβλεπτες καταστάσεις στην περίοδο εφαρμογής. Τώρα, να επανέλθω λίγο στο θέμα του περιθωρίου απρόβλεπτων. Mars pour l'imprevu. Η κυρία Ρούμπιο προτείνει να μην υπάρξει αργότερα αντιστάθμιση από αντίστοιχε περικοπές. Αυτό ήταν μια δυνατότητα για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, 2007 με 2009. Ήταν πολύτιμο, ναι, και το πέτυχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Διοργανική Συμφωνία και χρησιμοποιήθηκε μία φορά για την αναθεώρηση όσον αφορά τον Καλλιλέο το 2007, που ήταν η μόνη αναθεώρηση, ιστορικά μιλώντας, που εγκρίθηκε ποτέ με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο με μία χώρα μέλος κατά. Αλλά φοβάμαι ότι είχαμε την ε, συνθήκη της Λισαβόνας, συζητήσαμε νομικά για την ερμηνεία της συνθήκης της Λισαβόνας, οπότε φοβάμαι πως το συμπέρασμα στο οποίο έχουμε καταλήξει είναι ότι δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα αυτή γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ότι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να εγκρίνεται ομόφωνα και το ίδιο μας λένε και οι νομικοί εμπειρογνώμονες, άρα και οποιαδήποτε αναθεώρηση και αυτή θα πρέπει να περάσει ομόφωνα. Άρα εγώ δεν βλέπω να μπορούμε να πάμε πίσω στην κατάσταση πριν τη Λισαβόνα. Πριν ολοκληρώσω μια παρατήρηση ακόμα σχετικά με αυτά που λέει η κυρία Ρούμπιο γίνεται μνήα στην Επιτροπή λέγοντας ότι προτιμάει τη λύση 5 συν 5 για τη διάρκεια. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει παρεξήγηση. Η Επιτροπή δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι τώρα επ' αυτού και εξετάζει εξίσου όλες τις ε, δυνατότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φιντά. Κυρία Ρούμπιο. δεν ανέφερε νωρίτερα το ίδρυμα που εκπροσωπείται. Είναι το ίδρυμα Delor Ινστιτούτο Delor Notre Europe. Αν έχετε την καλοσύνη μπορείτε να απαντήσετε σε διάφορες παρατηρήσεις και θα δώσω το λόγο στο τέλος στο Γιάννου Ουλμπριχτ ε, για να απαντήσει, να κάνει τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Κυρία Ρούμπιο. Η κυρία Ρούμπιο, κύριε Ουλμπριχτ και μετά. Σας ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις και μερικές μάλιστα είναι άσχετες ε, με την ευελιξία και πολλές αφορούν περισσότερο το Brexit. Δεν θα επισέλθω στις λεπτομέρειες για το ποιες θα είναι οι συνέπειες ακριβώς του Brexit στον προϋπολογισμό. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σημεία που αφορούν ε, τη δική μου έκθεση. Ε, ε, η ανάγκη της μείωσης του προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής και της κοινής γεωρικής πολιτικής το χρηματοδοτικό κενό που θα αφήσει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου ε, θα είναι τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια το χρόνο, καθόλου αμεληταίο. Και αν το συγκρίνουμε το, το, σύνολο του κοινοτικού προπολογισμού, βλέπουμε ότι αφορά ένα σημαντικό ποσοστό. Είχαμε μια γραφική παράσταση που συγκρίναμε αυτό το χρηματοδοτικό κενό από τι διαφορέ ε, που υπάρχουν σήμερα και είναι πάνω από τον προπολογισμό του, του ορίζοντα 2020, 20% τη πολιτική συνοχή, 20% τη κοινή γεωργική πολιτική, ένα μεγάλο ποσοστό λοιπόν θα, των πολιτικών μας θα επηρεαστεί από αυτό το χρηματοδοτικό κενό και δεδομένη της σημασίας αυτού του κενού ε, δύσκολο θα μπορούμε να το αντισταθμίσουμε. Αν δούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το κενό, το χρηματοδοτικό ε, και πιστεύετε ότι θα το γεφυρώσουμε μόνο με την αύξηση των ιδίων πόρων, είναι μία πιθανότητα και αυτό αλλά πολιτικά θα είναι πολύ δύσκολο να εγκριθεί. Πολλό δε μάλλον όταν δεν υπάρχει αρκετό διάστημα για να θεσπιστούν νέοι ήδη οι πόροι. Επίσης η αύξηση των εθνικών συνεισφορών ε, θα είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτή από μερικά κράτη-μέλη. Οπότε χωρίς αύξηση εθνικών συνεισφορών, επίσης δεν μπορούμε να γεφυρώσουμε το κενό. Η μόνη λύση που βλέπω είναι να μειωθούν ε, οι προπολογισμοί των ε, δύο μιζώνων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, της συνοχής και της γεωργικής πολιτικής. Γιατί αν διασφαλίσουμε άθεκτο τους προπολογισμού στη συνοχή και στη γεωργική πολιτική θα πρέπει να περικόψουμε άλλες πολιτικές. Οπότε ούτως ή άλλως θα χρειαστεί μια ανακατανομή και των κονδυλίων μεταξύ των πολιτικών προτεραιοτήτων. Ε, ναι, και αν αναγνωρίσουμε σε ένα σενάριο ότι είναι σημαντικές παρόλα αυτά οι δύο πολιτικές ε, συνοχής και γεωργίας θα πρέπει ε, να συμφωνήσει φυσικά και το Συμβούλιο αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα αποκλείεται να μην περικοπεί καθόλου ο προπολογισμό τους. Τώρα, ε, ποιο θα είναι το ύψος του λογαριασμού που θα πληρώσει το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό είναι μια εκρεμή συζήτηση. Πάντως για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό αυτός ο λογαριασμός του Brexit να μην επιδεινώσει το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τα υπόλοιπα προς τα εκκρεμή από το τρέχον πι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αλλιώ θα χρειαστούν περισσότερε πιστώσει πληρωμών στο επόμενο πολίτε δημοσιονομικό πλαίσιο, άρα πολύ περισσότερα προβλήματα για το επόμενο πολίτε δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίση όταν μιλούμε για το μέγεθο του πι του επόμενου, ε, πολλά ακούμε για την ε, αύξηση του σχετικού μεγέθους του πι. Ωραία, πολύ ωραία. Αλλά άσχετα με το τι θα γίνει με το χρηματοδοτικό κενό του Brexit, θα έχουμε ούτως ή άλλως σε σχετικούς όρους μείωση, γιατί μια και η Βρετανική οικονομία είναι μεγάλο τμήμα του ποσοστού της ευρωπαϊκής οικονομίας, ακόμη και αν καλύψουμε το χρηματοδοτικό κενό και αυξήσουμε ή κρατήσουμε μετάβλητες τις δαπάνες, Παρόλα αυτά, ο κοινοτικό προπολογισμό σε σχετικού όρου θα μειωθεί. Είναι αδύνατο να κρατήσουμε τον προπολογισμό στο 1%. Γιατί ούτω ή άλλω θα φτωχύνει κατά κάποιο τρόπο η ευρωπαϊκή οικονομία με τον Brexit. Και ακόμη και αν σε σχετικούς όρου οι δαπάνε αυξηθούν, σε ουσιαστικούς όρου θα μειωθούν. Γιατί με το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα έχουμε πολύ μεγαλύτερο κοινοτικό προϋπολογισμό σε πραγματικούς όρους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ευελιξία. Όταν μιλούμε για την ευελιξία, αυτό που θα πρέπει να σας προβληματίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι έχουμε δύο τρόπους να το αντιμετωπίσουμε. Συμπληρωματικούς, δεν αλληλοαποκλείονται. Μπορούμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε τα, τις διατάξεις και τους μηχανισμούς ευελιξίας ή μπορούμε να αναθεωρήσουμε κάποια μηχανισμούς ευελιξίας, να τους δεχτούμε ή όχι, να αναθεωρήσουμε μερικούς, να τροποποιήσουμε τη διάρκεια ή τη δομή του ΠΔΠ και ο συγχρονισμός είναι πολύ σημαντικός, να συγχρονίσουμε το ΠΔΕΛΤΑΠ με τις πολιτικές εντολές, δηλαδή τις, την κοινοβουλευτική θητή, τη θητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη θητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αν ε, δούμε το συνολικό περιθώριο για τις υποχρεώσεις, περισσότερο χρησιμοποιήθηκε για να προσαρμοστούμε στις νέες προτεραιότητες της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε δράση και τα καθήκοντά της ένα χρόνο μετά την θέση εφαρμογή του νέου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Οπότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στη νέα Επιτροπή την ικανότητα να συμπεριλάβει στο ΠΔΕΛΤΑΠ και τις δικές της ε, δημοσιονομικές προτεραιότητες. Και το ίδιο ισχύει και για το Συμβούλιο και, την Επιτροπή, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό και χρειάζεται σημαντική ευελιξία. Αν το ΠΔΠ δεν συγχρονίζεται με τις πολιτικές εντολές και τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, χρειαζόμαστε μεγάλη ευελιξία για να προσαρμοστούμε στις δημοσιονομικές προτεραιότητες των νέων οργάνων που αναλαμβάνουν, των νέων εντολών και για την αύξηση της ενίσχυση της ευελιξίας είτε θα έχουμε περισσότερα περιθώρια και καλύτερη χρήση τους ή θα δημιουργήσουμε μηχανισμούς εκτός του ΠΔΠ όπως είναι αυτοί οι δικοί μηχανισμοί. Και αυτό εξαρτάται και από τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενότητα του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και την ε, βούλησή τους μερικοί μηχανισμοί να εντάσσονται ή να εξαιρούνται από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ή να περιλάβουμε περισσότερη γενή ευελιξία στα προγράμματα δαπανών. Και εκεί έχουμε σημαντικό δυναμικό που δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη στο έπακρο. Συμφωνώ απόλυτα με το θέμα του Ταμείου Μετανάστευσης. Όταν βλέπουμε πώς λειτουργεί σήμερα το Ταμείο, διαπιστώνουμε ότι έχει γίνει προσημείωση σχεδόν όλων των κονδυλίων. Και σίγουρα η προσφυγική κρίση ήταν μία από τις σημαντικές κρίσεις που σαν ανάγκη ευελιξίας, ενώ το αντίστοιχο πρόγραμμα ήταν άκαμπτο. Και εκεί είδαμε την αντίφαση που υπήρχε ε, και τη δυσκολία μερικές φορές ε, να προγραμματίσουμε τόσο συγκεκριμένα εκ των προτέρων κάποιες ανάγκες που στο, στην πορεία θα αλλάξουν. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιάννου. Δεν θέλω να σας ε, κρατήσω περισσότερο σύντομες παρατηρήσεις σε σχέση με την παρουσίασή σας. Και πριν λάβω το λόγο οι συνάδελφοι, ήθελα να επισημάνω ότι ήταν ενδιαφέρον αυτό που είπατε προς το τέλος, ότι δεν σκοπεύετε να επισέλθετε σε μια ανάλυση του Brexit, διότι δεν αφορά την ευελιξία. Αλλά προτείνετε το, τις περικοπές στη συνοχή και στη γεωργία, που πάλι δεν είναι ευελιξία αλλαγή πολιτική είναι και δομή του προπολογισμού. Επομένως δεν πρόκειται για ευελιξία, πρόκειται για μια πολιτική πρόταση αλλαγή πολιτικής. Επίσης ενδιαφέρον μου φαίνεται το γεγονός ότι αναφέρεστε σε μεταβατικό πολιτικο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή συζητούμε τι θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Και επίσης στην πρότασή σας για τροποποίηση ενός από τα μέσα που προβλέπει, προ... που προβλέπει αντιστάθμιση, μας λέτε ότι δεν πρέπει να γίνει αντιστάθμιση. Μα δεν είναι το ίδιο μέσο όμως τότε, αν δεν έχει αντιστάθμιση. Αποθυματικό είναι. Και επίσης, ενίσχυση ειδικών μέσων εκτός του πουδουπού. Τι εννοείται εκεί. Θέλω να ακούσω και τι θα πει ο επόμενος ομιλητής. Είναι ενδιαφέρον που το θίγετε σας έτσι. Είπαν όμω και οι συνάδελφοι ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που συζητούμε, αυτό για το οποίο οργανιζόμαστε εξ αρχής, είναι ένα πιο ευέλικτο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εάν θέλουμε περισσότερη ευελιξία, πρέπει να δούμε τι είδους ευελιξία θέλουμε. Θέλουμε ευελιξία Αυτή που προετοιμάσουμε εδώ και καιρό με την προετοιμασία και την κατάρτιση του Πουδουπού και των προτεραιοτήτων του για το Πουδουπού δεν είναι μόνο χρήμα, είναι πολιτικές. Θέλουμε να συζητούμε τις πολιτικές, θέλουμε ευελιξία για μια αιτία έτσι ώστε να μπορούμε να αλλάζουμε, να μετακινούμε ή να μετακινούμαστε μεταξύ προτεραιοτήτων όταν σε μια χρονική στιγμή όπως και τώρα. Άλλωστε δεν μπορούμε να προβλέπουμε ότι αφού έχει εγκριθεί το πουδουπού έρχεται η Επιτροπή και καταθέτει νέα προγράμματα. Τα οποία μπαίνουν στο χώρο της ε, ευελιξίας που δεν έχει προγραμματιστεί για τα νέα στοιχεία αλλά για τα υφιστάμενα στοιχεία. Επομένως, να κάποιο έρχεται με νέε ιδέες, νέα προγράμματα, πρέπει να δώσει και νέο χρήμα. Αλλιώ παίρνουμε το χρήμα της ευελιξίας που ήταν για τα ήδη ισχύοντα. Κάπω το λέτε και αυτό. Και γι' αυτό όταν ε, μιλούμε για ευελιξία και είναι ενδιαφέρον βέβαια για του συναδέλφου αυτό Ότι δηλαδή το που πρέπει να δίνει διαφορετικές λύσεις για την ίδια πολιτική, αλλά όταν παίρνουμε αποφάσεις για την ε, πολιτική που θα επιδιώξουμε, πρέπει να έχουμε ένα περιθώριο κινητικότητας επειδή οι συνθήκες αλλάζουν. Ακόμα και αν τρέχει ένα πρόγραμμα, αλλάζουν οι συνθήκες, άρα χρειάζεται περισσότερη ευελιξία. Αλλά η ευελιξία είναι απαραίτητη στο πουδουπού ή στον ετήσιο προπολογισμό γιατί στον ετήσιο προπολογισμό θα θέλαμε να απορροφώνται όλα τα κονδύλια, να τα δαπανούμε. Δηλαδή δεν θέλουμε περισσότερα αποθεματικά στο τέλος. Το είπε και ο Ζωζέ. Το Συμβούλιο θα είναι πολύ ευχαριστημένο αν δεν εκτελούμε τον προπολογισμό πλήρως κάθε έτος. Είναι μια φιλοσοφική επιλογή. Εμείς δεν θέλουμε να υποεκτελεί το προπολογισμό, θέλουμε να εκτελείται κατά το μέγιστο δυνατό, αλλά με τη δυνατότητα, την ευελιξία να κάνουμε μια διόρθωση και όχι τα αποθυματικά να τα αξιοποιούμε για τελείω νέε ιδέες. Δεν θέλουμε να βρεθούμε κάποια στιγμή να έχουμε αποφασίσει το πουδουπού και μετά, ένα χρόνο μετά την απόφαση να εμφανιστεί κάποιο να πει Α, έχω μια τελείω καινούργια ιδέα. Ελάτε να την ε, υλοποιήσουμε. Και να πάρω και ένα κομμάτι από τα χρήματα του πουδουπού. Το περιγράψατε κάπως, το βρήκα ενδιαφέρον. Και για να ολοκληρώσω, συνοψίζοντας, δεν αποφύγατε την ε, συζήτηση του ίδιου του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, όπως και εμείς. Δεν αποφασίζουμε εμείς το Brexit δεν αποφασίσαμε εμείς το Brexit, το, αποφασίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να το αποδεσμεύσουμε από τα υπόλοιπα. Είναι όλα λιλίνδετα μεταξύ τους. Και άρα το επιχείρημα που μας προσφέρεται είναι ότι πρέπει και να διαφυλάξουμε την διαφανή αλλά και να την καταστήσουμε στο δυνατόν πιο απλή και διαφανή γίνεται την ευελιξία. Αλλά θα ήθελα να ακούσω και τι άλλα ειδικά μέσα υπάρχουν. Την επόμενη δηλαδή παρουσίαση. Εκτός του πολίτου δημοσιονομικού πλησίου. Θα επικυρώσετε αυτά που είπε η κυρία Ρούμπιο ή θα μας προτείνετε κάτι τελείως διαφορετικό. Ο πρόεδρος ευχαριστώ. με διευκολύνεται κιόλα, ακριβώς το λόγο έχει τώρα για τον ενίο προπολογισμό, το πολιτισμικο δημοσιονομικό πλαίσιο και τον ενίο προπολογισμό, ο κύριος Μπέκερ από την Επιτροπή των προπολογισμών. Έχετε το λόγο κύριε Μπέκερ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Είναι τιμή για μένα. Συγγνώμη, είμαι κρυωμένο και ελπίζω εσεί και οι διερμηνεί κυρίω να καταφέρετε να καταλάβετε τι λέω, γιατί η φωνή μου είναι κάπω αλλοιωμένη. Θα αρχίσω με γενικέ παρατηρήσει. Ω γενική εισαγωγή για τι διαπραγματεύσει όσον αφορά το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και θα ε, καταλήξω και σε κάποια μαθήματα από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις και μετά θα έρθω στα πιο ειδικά θέματα που είναι η ενότητα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και τα άλλα που με ρωτήσατε για τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Ένα διαφορετικό προϋπολογισμό για την Ευρωζώνη δηλαδή. Λοιπόν, είναι ίσως μικρά εδώ τα γράμματα, αλλά έχετε και τα χαρτιά μπροστά σας νομίζω. Το σύστημα, όπως γνωρίζουμε σήμερα, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, 30 χρόνια αυξήθηκε και μετά βρέθηκε σε status quo με περιορισμούς ανάλογα με τα εθνικά συμφέροντα των χωρών μελών. Υπήρξε η δίκαια επιστροφή, το του ρετούρ», και μεταρρυθμίσεις που έγιναν με διάφορα μικρά βήματα. Όταν λοιπόν κοιτάξουμε την εμπειρία που έχουμε μέχρι τώρα, φαίνεται εδώ από τις διαπραγματεύσεις, καταλήγουμε να δούμε τι γινόταν με τα πακέτα του προπολογισμού στα τέλη της δεκαετίας 80, και της δεκαετίας 90, Delor 1, Delor 2, που ήταν δύο πακέτα τότε και Σχετικά με αυτό μπορούμε να κάνουμε τρεις παρατηρήσεις. Να δούμε πόσο κράτησε η διαδικασία διαπραγματεύσεων προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία μεταξύ των χωρών μελών και να καταλήξουμε σε συμβιβασμό μεταξύ των χωρών μελών Επιτροπή και Συμβούλιο. Από 12 μήνες σε σχεδόν δύο χρόνια βλέπουμε ότι κρατάνε διαπραγματεύσεις αυτές. Έπειτα απόλυτα αυξήθηκε ο προπολογισμό. Σχετικά όμως, δηλαδή σε σχέση με το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώθηκε ο προπολογισμό. Και η τρίτη παρατήρηση, τη βλέπετε στην τελευταία στήλη, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα προσπαθεί να συνδυάσει την πρότασή της με ένα κοινό ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να πει σε όλες τις χώρες μέλη δηλαδή στις διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ότι χρειάζονται περισσότερα ποσά για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, για παράδειγμα για τη διεύρυνση το 2000 κλπ θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πέτυχε να συνδυάσει το παλιό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το επόμενο, με τα μετά τη Λισαβόνα. Θα έλεγα ότι δεν ήταν πιστική ούτε απέναντι στο Συμβούλιο. Τι διδάγματα μπορούμε να πάρουμε. Πρώτον, ότι οι διαπραγματεύσεις ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση και αλλαγή παίρνουν χρόνο, πολύ χρόνο για να φτάσουμε σε συμβιβασμό. Και αν συμπεριλάβετε και τις νομικές επιπτώσεις των δημοσιονομικών συμβιβασμών στις διάφορες πολιτικές ε, από τις οποίες χρησιμοποιούμε κονδύλια και αυτό είναι χρονοβόρο. Το δεύτερο είναι από την εμπειρία αυτή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να βρει και να αναπτύξει μια νέα πιστική ιδέα. Με ένα επιχείρημα ευρωπαϊκό για να πείσει και τις χώρες μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η μεταρρύθμιση της δημοσιονομικής πολιτικής είναι αναγκαία. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει προθυμία στη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ο κόσμος προτιμάει να χρησιμοποιεί αυτά που γνωρίζει, ακόμα και γνωρίζει και τις αδυναμίες τους. Οπότε, το μόνο που μπορεί να ενώσει τις διαπραγματεύσεις όλους τους παίκτες είναι ότι στο τέλος, έτσι κι πρέπει να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς. Είναι πιο σημαντικό, αυτό δηλαδή πρέπει να πιστούν, ότι είναι πιο σημαντικό να έχουμε ένα νέο νέο πολιτισμο-οικονομικό πλαίσιο παρά να κάνουμε διορθώσει δεξιά και αριστερά στα παλιά. Συνεπώ, διαπραγματεύσει είναι δύσκολε και για μένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να τονίσει την προστιθέμενη αξία. Και αυτό να υπερισχύσει μετά το 2020. Όμω, υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί για το τι θα μπορούσε να είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και πώς μετράται αυτή. Περισσότερη αποτελεσματικότητα, ε, συσχετισμός κόστους κόστους-οφέλους, ε, ε, δομές, ε, συνεργασίες. Άλλοι λένε είναι τα ταμεία συνοχής, η γεωργική πολιτική, εκεί δηλαδή που ξοδεύεται ευρωπαϊκό χρήμα για ένα σκοπό. Δεν υπάρχει λοιπόν κοινό ορισμό για το τι είναι αυτή η προστιθέμενη αξία. Και ενώ παραδοσιακά η πρώτη πράξη στις διαπραγματεύσεις ήταν και είναι να προσπαθήσουμε να πετύχουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα και να βρούμε αυτή την προστιθέμενη αξία και όλες οι χώρες μέλη, όλες οι πλευρές συμφωνούν με την αρχή αυτή, Τελικά, αυτή η αρχή μπαίνει κάπως ε, στην πάντα και μιλάμε πιο πολύ για πολιτικές από τις οποίες ε, ξοδεύουμε χρήματα. Οπότε μένει ανοιχτό αυτός ο ορισμός. Το άλλο είναι τώρα πώς θα δαπανίσουμε αποτελεσματικά τα χρήματα των φορολογούμενων που έτσι κι αλλιώς δεν είναι άπειρα. Σε αυτό καταλήγουμε στο τέλος των διαπραγματεύσεων. Οπότε, οι διαπραγματεύσεις μερικές φορές σε κάποια σημεία γίνονται επιφανειακά. Θέλω να πω ότι αυτή η έννοια της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσει να τραβήξει όλο το κόσμο και να φροντίσει όλος ο κόσμος να σταθεί σε αυτό και αυτό να θελήσουν όλοι να προωθήσουν, γιατί ο καθένα καταλαβαίνει κάτι διαφορετικό γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, θα έπρεπε στι διαπραγματεύσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο να βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι στο τέλο. Πάμε παρακάτω. Ας δούμε τώρα πώς διαρθρώνονται οι διαπραγματεύσεις. Συνήθως, για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ξέρουμε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις κάθε φορά είναι πιο δύσκολες από τις προηγούμενες. Πάντα η επόμενη διαπραγμάτευση είναι η πιο δύσκολη. Όμως αυτή τη φορά ισχύει. Θα έχουμε νέες προκλήσεις, Brexit, το συζητήσαμε ήδη, εξαιτίας της κρίσης στην Ευρωζώνη που πρέπει ακόμα να αντιμετωπιστεί και εξαιτία των προσδοκιών για περισσότερη κοινωνική Ευρώπη, για περισσότερη ασφάλεια στην Ευρώπη. Άρα υπάρχουν προσδοκίες για επιπλέον αρμοδιότητες και άρα επιπλέον χρηματοδότηση. Καλά, δεν θα μιλήσουμε για το Brexit, ε, διπλό κενό Brexit στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι όσοι χώρες δεν γνωρίζουν αυτό το κενό από το Brexit θα είναι, και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται από αυτού, για το οικονομικό κενό δηλαδή, δύσκολα οι χώρες μέλη μπορούν να διαπραγματευτούν για χρηματοδότηση νέων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, γιατί δεν ξέρουν τι χρήματα θα έχουν στη διάθεσή τους. Και τι χρήματα θα μπουν στον ευρωπαϊκό κορβανά. Μια άλλη πρόκληση για τις διαπραγματεύσεις είναι το χρονοδιάγραμμα, που είναι και αυτό πολύ δύσκολο αυτή τη φορά. Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2019 ή αρχές του 2020 αν θέλετε να μπορέσετε να προετοιμάσετε καλά τα πολυετή προγράμματα. Η Γεωργία, ο Ορίζοντας 2020, Post 2020 κλπ. Αν όμως οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, τότε το χρονοδιάγραμμα θα έχει ω εξή. Η Επιτροπή θα υποβάλει την πρότασή τη πριν τι καλοκαιρινέ διακοπέ του χρόνου, το Μάιο α πούμε, και τον Οκτώβριο τη επόμενη χρονιά την νομοθετική πρόταση για τα κονδύλια για την γεωργική πολιτική κλπ. Στη συνέχεια οι χώρες μέλη θα αρχίσουν να εξετάζουν συνολικά την πρόταση στην αρχή και μετά το δεύτερο ο του 2018 η Προεδρία εκεί θα αρχίσει να κάνει τις διαπραγματεύσεις κομμάτι-κομμάτι και μετά το πρώτο εξάμεινο του 2019 Ρουμανική Προεδρία. Και αν δεν υπάρχει αρκετή συνένεση στο Συμβούλιο, τότε θα πρέπει στο Συμβούλιο να γίνουν διαπραγματεύσεις και μετά το 2019 θα περάσουμε στις ε, τελικές. Ε, συνήθως δύο προσπάθειες γίνονται μέχρι να πετύχουμε. Η πρώτη είναι, ας πούμε, για τα μάτια του κόσμου, τέλο πάντων, για να εκφράσει ο καθένας τα δικά του συμφέροντα και να προσπαθήσει τέλο πάντων ό,τι μπορεί να κερδίσει, να κερδίσει. Και τη δεύτερη φορά είναι που τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά. Μετά τώρα τις εκλογές του 2019 θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, δηλαδή το φθινόπωρο του 2019. Και θα έχουμε ένα νέο κανονισμό μετά την Άνοιξη του 2020. Εφόσον λοιπόν έχει έτσι το χρονοδιάγραμμα, η προετοιμασία για μετά το 2020, η περίοδος θα είναι πάρα πολύ μικρή. Και συγχρόνως θα έχουμε και τις τελικές διαπραγματεύσεις για το Brexit και θα δείτε να λήγουν και η εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Επιτροπής που σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για το Πουδουπού θα γίνουν συγχρόνως με εκλογές, με επιλογή ε, των ε, αξιωματούχων στην τράπεζα, επιτροπή και τα με επιλογή νέου προσωπικού, που ίσως όλα αυτά όπως και το Brexit να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και πρέπει να δούμε κατά πόσο τόσο θα μπορέσει, θα, το επιτρέψει μια χώρα μέλο να ε, διαπραγματευτεί στο Συμβούλιο την τελική συμφωνία. Όλα αυτά γίνονται πολύ περίπλοκα για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Άρα έχουμε ένα περίπλοκο χρονοδιάγραμμα με νέες προκλήσεις σε ένα δύσκολο περιβάλλον και με χρονικούς περιορισμούς. Τώρα για την δημοσιονομική ενότητα. Η συμμετοχή και ο έλεγχος είναι προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη δημοσιονομική πολιτική και συνδέονται με τον προπολογισμό. Το ότι είναι ενιαίο ο προπολογισμό, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό και συνδεδεμένο άρρητα με τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Όπω όμω είπαμε, υπάρχουν κάποιε δυνατέ εξαιρέσει και αναγκαίε μάλιστα από αυτήν την αρχή του ενιαίου προπολογισμού. Όπω είναι το αναπραξιακό ταμείο ε, πράγματα τα οποία αναφέρονται στο πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο. Σήμερα μπορούμε να συνοψίσουμε πάντως ως εξής. Υπάρχει μεγάλος κατακερματισμός μέσων εργαλείων και μέσα στον προπολογισμό και εκτός. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, τα διάφορα καταπιστεύματα, τα trust funds, γιατί είναι εκτός προπολογισμού όλοι αυτοί οι μηχανισμοί και τα εργαλεία. Θεωρήθηκε αναγκαίο για να μπορούμε να έχουμε κάτι ελαστικό, ευέλικτο, που να μας επιτρέπει πιο εύκολα να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Αυτό είναι ένας λόγος και άλλος είναι ότι έτσι έχουμε νέο χρήμα. Χωρίς να χρειάζεται να περάσουμε από διαπραγματεύσεις και να αλλάξουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχει τάση, ένα παζάρι τέλος πάντων ε, που γίνεται ανάμεσα στην ευελιξία και τον μακροχρόνιο σχεδιασμό. Πάντως το αποτέλεσμα από την ευελιξία και την ταχύτητα με την οποία θέλουμε να λαμβάνουμε αποφάσεις είναι πρώτον ότι τα προνόμια του Κοινοβουλίου απέναντι στον προπολογισμό βράχει κυκλώνονται κάπως. Έτσι, ναι, μεν οι αποφάσεις λαμβάνονται πιο γρήγορα από τις χώρες μέλη και την Επιτροπή, αλλά όχι με περισσότερη νομιμότητα από την άλλη. Δεύτερον, για τον προελθό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εθνικούς προπολογισμούς μπλέκονται μεταξύ τους για να χρηματοδοτηθεί το ένα ή το άλλο πρόγραμμα. Τρίτον, τα νέα μέσα δίνουν μια πολιτική ευχαίρεια εφόσον φέρνουν νέο χρήμα, αλλά το δημοσιονομικό σύστημα του προπλογισμού γίνεται πιο περίπλοκο και χάνουμε σε διαφάνεια. Εδώ βλέπετε κάποια αξιολόγηση κατά κάποιο τρόπο του κοινοβουλευτικού έργου για έλεγχο, απαλλαγή των ε, των μηχανισμών αυτών και των ε, χρηματοπιστωτικών μέσων που βρίσκονται εκτός προπολογισμού. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια ταξινόμηση, μια ιεράρχηση. Πώς να ιεραρχήσουμε αυτά τα μέσα, εντός ή εκτός προπολογισμού και πώς έχει η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάθε φορά. Είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα που θα έπρεπε να αναλυθεί και γίνεται. Με τον πίνακα αυτό έχετε κάποια ιδέα για το πώς θα έπρεπε να είχε μια τέτοια ταξινόμηση, μια ιεράρχηση, συνδέοντας τη συμμετοχή, τη δυνατότητα συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όχι, με την χρήση κοινοτικών κονδυλίων Νομίζω ότι έχουμε ακρηγορήσει, Πρόεδρε, έτσι. Κοιτάω λίγο ανήσυχο στο ρολόι μου, όπως βλέπετε. Έχετε δίκιο, λοιπόν, αν μπορείτε να ολοκληρώσετε. Μια πρόταση ακόμα, επιτρέψτε μου. Για το θέμα του προπολογισμού της Ευρωζώνης, που είναι μια ειδική περίπτωση διαφοροποίησης και κατακαιρματισμού του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Είναι ανοιχτό ακόμα το ζήτημα και οι συνέπειες είναι διαφορετικές για το ενίο του προπολογισμού. Πώς αποφασίζεται αυτός ο προπολογισμό τη Ευρωζώνη. Πάντως για να επανέλθω στο κεντρικό ζήτημα, μέσα ή έξω από τον κοινοτικό προπολογισμό, αυτού του προπολογισμού για την Ευρωζώνη, να ξέρετε ότι υπάρχουν παραδείγματα και υπάρχουν τρόποι να δημιουργηθεί ο προπολογισμό αυτό ε, τη Ευρωζώνη μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αν θέλετε να δημιουργήσετε αυτήν τη δημοσιονομική ικανότητα, το πάντων αυτό το προπολογισμό Ευρωζώνης εκτός προπολογισμού, με διαφορετική διακυβέρνηση, ε, υπουργό για την Ευρωζώνη, τότε αυτό ίσως σημαίνει ότι μπορεί να γίνει πιο εύκολα και να είναι πιο εύκολο να διαπραγματευτούν μεταξύ τους οι χώρες για έναν τέτοιο προϋπολογισμό ευρωζώνης. Αλλά έτσι ενισχύεται ο κατακαιρματισμός και χάνεται ο ενίος χαρακτήρας του κοινοτικού προϋπολογισμού και της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Δόκτωρ Μπέκερ κύριος Κρόους. Κρίτσαρτ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Θα εξετάσουμε τώρα το θέμα και από πιο νομική πλευρά. Από νομική απόψεω, το σημείο αναφοράς μας είναι η συνθήκη της Λισαβόνα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι οι δημοσιονομικές διατάξει της συνθήκης της Λισαβόνα ε, εκπονήθηκαν στη συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης, ε, που έγινε το 2002-2003 εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και οι δημοσιονομικές διατάξεις ε, ε, προήλθαν από την ομάδα εργασίας για την απλούστευση. Και αν θυμάστε τα έγγραφα που είχαν κυκλοφορήσει τότε από τη συντακτική συνέλευση, θα διαπιστώσετε ότι στόχος ήταν να γίνει το σύστημα σαφέστερο και πιο κατανοητό για τους Ευρωπαίους πολίτες και να είναι σαφές ποιος κάνει τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ε, δούμε όμως τι συνέβη από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο κατακαιρματισμένα και πιο περίπλοκα. Καταρχήν, στο πλαίσιο ε, της χρηματοπιστωτικής ε, και κρίσης του δημόσιου χρέους, ε, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, διαχείριση μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης. Έχουμε όλο και μεγαλύτερη χρήση αυτών των υβριδικών μέσων που λέμε, δηλαδή συνδυασμό του κοινοτικού προϋπολογισμού με τις κάποια μέσα που συνεισφέρουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί. Το άρθρο 310 παράγραφος 1 της συνθήκης προβλέπει και κατοχυρώνει την αρχή της ενότητας, δηλαδή όλα τα έσοδα και έξοδα της Ένωσης θα πρέπει να εφαίνονται στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Βέβαια η συνθήκη προβλέπει και τη χρηματοδότηση κάποιων προηλητικών από τα κράτη-μέλη άμεσα, όπως η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, ενισχυμένη συνεργασία. Εδώ καταρχήν έχουμε ε, χρηματοδότηση και συμμετοχή των κρατών μελών. Βέβαια, έχουν γίνει κάποιες παραβιάσεις της αρχές της ενότητας. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει ότι μηχανισμοί όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Σταθερότητας που χρησιμοποιούν θεσμικά όργανα, την, την Επιτροπή, το ΕΚΤ, ε, και χρησιμοποιούν και μέσα, θεσμικά όργανα εκτός της συνθήκης είναι συμβατά. Αυτή ήταν μια σχετική νομολογία. Ο, εξού και ο κατακαιρματισμός που έχει προκύψει. Είναι αντίθετος με τις συνθήκες, όχι γιατί υπάρχει και νομική βάση γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά συμβάλλει αυτός ο κατακαιρματισμός στη μεγαλύτερη περιπλοκότητα και αντιβαίνει στον αρχικό στόχο της Ένωσης που ήταν ένας απλός και κατανοητός προϋπολογισμός για τους πολίτες που θα γνωρίζουν ποιος κάνει τι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και φυσικά κάτι τέτοιο έχει επιπτώσεις και για το κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Σε κάποιο βαθμό τα μέσα της Ευρωζώνης όπως ο ESM είναι ε, μηχανισμοί που ακολουθούν ε, το το ιστορικό που είδαμε προηγουμένω και με τι κρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλήφθηκε ότι θα πρέπει να κάνει κάτι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, για πολλού και διάφορου λόγου γίνεται τέτοιο αρχικά σε διακυβερνητικό επίπεδο και κατόπιν συμπεριλαμβάνεται τα μέτρα αυτά ε, στη συνθήκη. Είδαμε τι έγινε με, τη εσωτερικέ με τις εσωτερικές υποθέσεις ε, και τη συνθήκη του Μάστριχτ. Αρχικά ε, μπήκαν κάποιες, ε, έγιναν κάποιες αποφάσεις διακυβερνικά και στη συνέχεια σωματώθηκαν στην συνθήκη. Τώρα για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα έχουμε μια πιο μακροχρόνια μεταβατική περίοδο, αλλά μακροπρόθεσμα θα συμπεριληφθούν και τέτοια μέτρα και μηχανισμοί στο πλαίσιο της, των συνθήκων. Τώρα, ε, είδαμε στο τελευταίο πι ε, τη χρήση κάποιων υβριδικών ε, μέσων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνδυασμό κοινοτικών κονδυλίων και κρατικών κονδυλίων για να παρακάμψουμε τα ανώτατα όρια των ΠΙΔΕΛΤΑΠ, για παράδειγμα, η διευκόλυνση για τους πρόσφυγες ε, στη συμφωνία με την Τουρκία. Τώρα, επανέρχομαι στο, στη συνθήκη της Λισαβόνας και το στόχο της απλούστευσης. Ε, σε κάποιο βαθμό παρά ήταν απλουστευτική η συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, αναφέρθηκε μάλιστα ότι το ΠΔΠ θα κατοχυρώνεται σε κανονισμό με ανώτατα όρια και ο κανονισμό θα πρέπει να εγκρίνεται με ομοφωνία. Πολύ ωραία όλα αυτά, να βάζουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ξεκάθαρα στη συνθήκη και σε ένα κανονισμό, αλλά ο κανονισμός είναι ένα πολύ απότομο ε, νομικό εργαλείο. Προηγουμένω είχαμε τη διοργανική συμφωνία, που είναι πολύ πιο ευέλικτο εργαλείο και μπορεί να τροποποιείται πιο απρά. Τώρα έχουμε κανονισμό και από τη θέση τη συνθήκη τη Λισαβόνα, ο κανονισμό για το ΠΔΠ έχει σχεδόν αποκτήσει την ε, ισχύ μια συνθήκη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέμε κάποιο έχει καλή ιδέα, αλλά του λέμε όχι δεν γίνεται να εφαρμοστεί γιατί απαιτείται μεταρρύθμιση της συνθήκης. Ε, ε, στα δημοσιονομικά ε, λέμε κάτι που θα μπορούσε καλό θα ήταν να γίνει, αλλά είναι αδύνατο, ανέφικτο, επειδή θα προϋπέθεται τροποποίηση του ΠΔΠ. Έχει δηλαδή ε, αποκτήσει το ΠΔΠ σχεδόν αξία συνθήκης. Τώρα, το, η συνθήκη προβλέπει κανονισμό για το ΠΔΠ. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Καταρχήν να διδαχτούμε τα, από τα παθήματα του τελευταίου ΠΔΠ και να έχουμε υψηλότερα ανώτατα όρια. Επίσης, ε, να ενισχύσουμε τους ειδικούς μηχανισμούς εκτός του ΠΔΠ. Λέμε, δεν θα χρειαστεί γιατί θα είναι αρκετά τα ανώτατα όρια. Επίσης, η βάση για τους ειδικούς μηχανισμούς προτείνεται στο άρθρο 322 παράγραφος 3 Εκεί αναφέρονται ότι το ΠΔΠ θα περιλαμβάνει ανώτατα όρια και ε, τις απαραίτητες διατάξεις για να επιτρέψουν την εύρυθμη διεξαγωγή της ε, ετήσιας δημοσιονομικής διαδικασίας. Οπότε προβλέπεται τέτοια ευελιξία στα πλαίσια του ετήσιου προπολογισμού. Και παρόλο που ο κανονισμός είναι πολύ ξεκάθαρο και ε, απότομο, κάπως άκαμπτο εργαλείο, υπάρχουν δυνατότητες ε, ευέλικτων μέτρων και εντός του κανονισμού. Το είδαμε στα συνολικά περιθώρια για τις υποχρεώσεις και για τις πληρωμές. Τώρα έχουμε ιδέα για την ε, νέα χρησιμοποίηση κάποιων κονδυλίων, όπως είχαμε στην, στο αποθεμα... ή την πρόταση για το αποθεματικό της κρίσης. Και ενώ αρχικά είχαμε πει ότι είναι αδύνατο ολικά περιθώρια για υποχρεώσει και πληρωμέ, είδαμε ότι τελικά γίνεται κάτι τέτοιο. Και μπορεί μια ιδέα αρχικά στην αρχή των διαπραγματεύσεων να απορριφθεί, αλλά μέχρι το τέλο να γίνει αποδεκτή. Σε ό,τι αφορά τη σαφή διατύπωση, αυτό αναφέρθηκε για τι πληρωμέ σε ειδικού μηχανισμού, αν θα είναι εντό ή εκτό των ανωτάτων ορίων. Την τελευταία φορά αντιληφθήκαμε το πρόβλημα, αλλά ήταν αδύνατο να συγκεντρώσουμε ομοφωνία ως προς τη σαφή διατύπωση εξού και η αόριστη διατύπωση μετακυλίωτας το πρόβλημα για την επόμενη επταετία. Κάποια στιγμή θα πρέπει να επανέλθουμε ώστε στην επόμενη συμφωνία η διατύπωση να είναι ξεκάθαρη και σαφής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, όλοι ο κύριος Γκαλιάς. Θα ήθελα για πρακτικούς λόγους ένα λεπτάκι να συνοηθούμε λίγο. Έχουμε συμφωνήσει ότι 5.30 θα, γίνει, θα ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες. Έχουμε επίσης ε, συμφωνήσει ότι θα έρθει και ο κύριος Πόνς για 30 λεπτά. Θα μας μιλήσει σε μια ανταλλαγή απόψεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη της Βιομηχανίας Άμυνας. Δηλαδή, στις 5 πρέπει να σταματήσει αυτό το κομμάτι των ε, συζητήσεων μας. 45 λεπτά μου λέει το ρολόι μου, μας μένουν ακόμη. Αν πιστεύετε και εσείς βέβαια ότι χρειάζεται με ακρίβεια και συγκέντρωση στη θεματολογία μας να προχωρήσουμε. Ας δούμε τώρα. Πρώτο είναι ο Γιάνν. Ολμπρίχτ. Εκπλήσουμε, δεν βλέπω τίποτα καινούριο ομολογώ, αλλά... έχω πράγματα που είμαστε συνηθισμένοι να ακούμε, ότι αφενός μεν δεν έχουμε ε, ενιαίο χαρακτήρα του προπολογισμού, δεν τον ελέγχουμε, δεν έχουμε το δημοκρατικό έλεγχο. Βρίσκεται όλο και περισσότερο εκτός κάθε δημοκρατικού ελέγχου ή εποπτείας από το Κοινοβούλιο. Αφενός, αφετέρου δε, απαιτείται περισσότερη ευελιξία, και αυτή η ευελιξία σημαίνει και ευέλικτα μέσα. Μια πρώτη παρατήρηση λοιπόν θα ήταν προς το κοινοβούλιο αφενός ερώτηση. Τι θέλετε, θέλετε την ευελιξία. Ευέλικτα μέσα τότε. Δεν θέλετε ευελιξία. Τότε μειώστε τα εξωτερικά μέσα. Και κονδύλια. Και ζητώ συγγνώμη που τα υπεραπροστεύω ίσως, αλλά πού θέλουμε να πάμε. Θέλουμε τα εξωτερικά κονδύλια και τα μία μέσα να είναι διπλάσια σε όγκο από τον προπολογισμό. Να έχουμε ένα μικρό προπολογισμό με διάφορα ε, δορυφορικά μέσα και ταμεία για να έχουμε την ευελιξία. Κάποια απόφαση πρέπει να πάρουμε. Τι παίζεται εδώ. Και υπερβάλλοντας πάντα, θέλετε ο προϋπολογισμός να μεταφραστεί σε ένα σύνολο μέσων, οπότε θα είναι τελείω διαφορετικό και ο έλεγχο με ένα διαφορετικό τύπο προπολογισμού ή θέλουμε έναν κύριο προπολογισμό με κάποια συμπληρωματικά μόνο μέσα και κονδύλια που ε, περιστρέφονται γύρω από αυτόν, αλλά είναι προσωρινά, προσωρινά μόνο για ένα διάστημα γιατί μετά ενσωματώνονται στον προπολογισμό. Διότι οι δάλωσαν, αν σταθεροποιηθούν και διατηρηθούν, θα διαρκήσουν για πάντα και θα είναι για πάντα εκτός του προϋπολογισμού όλο και περισσότερα μέσα κονδύλια ταμεία και έτσι δεν θα είμαστε ούτε καν στο 1 ή 1,24, στο 0,9, 0,8 και γύρω-γύρω θα είναι όλα τα εξωτερικά ταμεία. Τι θέλουμε, όχι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο πρέπει να ρωτήσουμε και το Κοινοβούλιο να πάρουν την απόφαση τι θέλουν. Γιατί έχετε απολύτω δίκαιο, εάν θέλετε το δεύτερο στοιχείο της ενότητας του προπολογισμού του προπολογισμού της Ευρωζώνης, αν είναι κάτι σαν Ιωνή προπολογισμό, ο προπολογισμό τη Ευρωζώνη, ή αν θέλουμε να ο προπολογισμό για την Ευρωζώνη. Είναι κάτι που επαναλημμένω έχει αναφερθεί ο πρώην Υπουργό των Οικονομικών τη Γερμανία, ο κ. Σόιμπλε. Τον θυμάμαι πολύ καλά. Πολλέ φορέ το έχει πει ότι χρειάζεται προπολογισμό τη Ευρωζώνη, προκοινοβούλιο τη Ευρωζώνη μάλιστα, που θα παρακολουθεί τις συνόδους ε, της Ευρωζώνης, μια νέα συνθήκη ευρώ κτλ. Τι θέλουμε όμως, τι θέλουμε αυτά, δεν μπορούμε να τα αποκρύψουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Απαντήσεις δεν δίνουμε, ε, μόνο ερωτήσεις προξενούν τα όσα μας είπε ο εμπειρογνώμων. Τι θέλετε και πώς θέλετε να δημορφωθεί όλη αυτή η κατάσταση. Είναι ενδιαφέρον το χρονοδιάγραμμα που παρακολουθεί τις εργασίες του Συμβουλίου. Μας και μετά τις εκλογές. Εμείς θα θέλαμε να είμαστε έτοιμοι πριν τις εκλογές. Το θέμα είναι να τα προλαβαίνουμε. Ή όπως είπε και η κυρία Ρούμπιο, περνάμε σε μεταβατικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό. Ευχαριστώ πάντως για τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα ως χαρτογράφηση. Βλέπουμε τι έχουμε γύρω μας. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι θέλουμε, που θέλουμε να πάμε και τι θα προτείνουμε. Γκάιερ. Ευχαριστώ. Μάλετιτς και μετά Μπούγκε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το υλικό που μας στείλατε και τις παρουσιάσεις που κάνατε. Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο Όλμπριχτ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας να έχουμε μια πολύ καλή και άρτια γενική επισκόπηση είναι ανεκτήμητης αξίας για να ετοιμαστούμε κατάλληλα. Στις ε, εκθέσεις που μας παρουσιάσατε ε, και στις διαφάνειες τονίσατε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ακόμη όμως αναζητούμε τον ορισμό της προστιθέμενης αξίας, της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και πώς θα καταμετρήσουμε αυτή την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Στην πολιτική συνοχή, για παράδειγμα, έχουμε θεσπίσει πολλές αρχές για να καταλήξουμε σε τελική ανάλυση στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Έξυπνη εξειδίκευση, θεματική συγκέντρωση, εκ των προτέρων ερεσιμότητα. Αλλά σε τελική ανάλυση το σύστημα με τις αρχές αυτές έχει γίνει τόσο περίπλοκο που πάλι στη τελική ανάλυση δεν έχουμε απόλυτη βεβαιότητα για το τι εστί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να πλουστεύσουμε τον τρόπο που καταμετρούμε αυτή την προστιθέμενη αξία, πώς την ποσοτικοποιούμε και να καθορίσουμε τη βασική αρχή, τη θεμελιώδη αρχή ε, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα αν κάτι όντως ε, ε, επιφέρει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Επίσης, σας ευχαριστώ για τις ιδέες που μας δώσατε για το χρονοδιάγραμμα. Ε, μιλήσατε για την άνοιξη του 2020. Νομίζω ότι είναι πολύ αργά άνοιξη του 2020. Αν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι στην πολιτική συνοχή στις αρχές του 2021, καλό θα ήταν όλα να έχουν διεκπαιρεωθεί στα τέλη του 2019 ώστε τα κράτη-μέλη να προετοιμαστούν και να ξεκινήσουν την εφαρμογή το 2021. Η δεμή θα έχουμε και πάλι καθυστερήσεις στις πληρωμές, όπως ε, πολύ σωστά μας παρουσίασε η κυρία Ρούμπιο, μια γραφική απεικόνηση όπου συγκρίνατε τις πληρωμές για, τη, για την περίοδο προγραμματισμού και την εκτέλεση στο 2007-2013 και μετά στο 2014 και 2014-2020 και είδαμε τις διαφορές με την εφαρμογή διαφορετικών αρχών. Αν θέλουμε λοιπόν να αποφύγουμε τέτοιες διαφορές μεταξύ προγραμματισμού και εκτέλεσης θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι πιο γρήγορα. Και το τελευταίο σχόλιο για το προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι ο η ύπαρξη ξεχωριστού προπολογισμού για την Ευρωζώνη θα επιτείνει τη διαφοροποίηση και τον κατακαιρματισμό του κοινοτικού προπολογισμού. Αν θέλουμε ένα προπολογισμό τη Ευρωζώνη, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ενταχθούν όλα τα κράτη-μέλη στην Ευρωζώνη. Και για να μπουν όλα τα κράτη-μέλη στην Ευρωζώνη, θα πρέπει να επιταχύνουμε την ουσιαστική σύγκληση για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να ενταχθούν στην Ευρωζώνη. Άρα θα πρέπει και πάλι να αυξήσουμε την πολιτική συνοχής, γιατί η πολιτική συνοχής ε, θα επιτρέψει ε, την μείωση των ανισοτήτων και την ε, ενίσχυση της σύγκλησης μεταξύ των κρατών μελών. Οπότε είναι σαφές ποιος θα πρέπει να είναι ο πρωταρχικός μας στόχος για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Πρόεδρε, ευχαριστώ. Παρακολούθησα την πολύ συναρπαστική αξιολόγηση της νομικής υπηρεσίας και σκέφτηκα ότι ναι, υπάρχουν αποφάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, του δικαστηρίου για, τις, ε, για τα ποσά, για τα κονδύλια και τα μία που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Πολυπροϋπολογισμού, ότι είναι σύμφωνα με τον, ε, Ευρω με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σύμφωνα, συμβατά, με ναι, αλλά όχι ε, επαρκώς διαφανή και βεβαίως είναι απαραίτητη για την πολιτική η διαφάνεια. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε και εδώ έχουμε την συζήτηση, είτε, πρόκειται για, είτε το λέμε ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, είτε άλλα μέτρα, ότι είναι φορές που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι άκρος δημιουργική και εφάνταστη ως προς τις ε, είναι στις νομικές. Βασικά, ό,τι τη βολεύει. Όπως όταν μπορέσαμε το 2009 να βρούμε δύο δις για να καλύψουμε τον προϋπολογισμό, για να ανακαλύψουμε μετά ότι υπήρχαν σοβαρά ζητήματα τουλάχιστον για εκείνους που όπως εγώ δεν είναι νομικοί. Ε, ρωτώ λοιπόν ποια είναι η κατάσταση τώρα. Το έθιξα και νωρίτερα. Σε ποιο πλαίσιο παραπέμπει σε συνθήκες η νομική υπηρεσία. Όταν είχαμε τη σταγματική συνέλευση, ο Τόμας Ζούμπελα πρόωρα απελθόν δυστυχώς, είχε πει τώρα οι κάτω χώρες βρίσκονται σε κρίση, οι ανώτατοι διπλωματικοί υπάλληλοι μέσα στο κτίριο του Κοινοβουλίου έρχονται να ε, Από διαρθρώσουν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ο κίνδυνος είναι τεράστιος, είναι σαν να πλημμυρίζουν οι κατοχώρες και έγιναν αμέσως διορθωτικές κινήσεις και προσαρμογές και νέα άρθρα και παράγραφοι έτσι ώστε όλοι να πούν ότι είμαστε τεθειμένοι να, δια... προσφέρουμε, να συνεισφέρουμε, να προσαρμόσουμε κτλ. Αυτό στις τελευταίες διαπραγματεύσεις του Πουδουπού και με το γεγονός ότι το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ομόφωνα μόνο άπαξ και έχει δώσει συνένες, ε, συμφωνία το Κοινοβούλιο, περίπλοκη διαδικασία το όντι. δόθηκε ένα περιθώριο κινητικότητας με επίκληση αυτής της παραγράφου για να μπορέσει και το Κοινοβούλιο να δει μια θετική κίνηση. Είπαμε όμως ότι θέλαμε να ενισχύσουμε περισσότερο τη διαδικασία, δηλαδή να είναι πιο ολοκληρωμένη, πιο ενοποιημένη αυτή η διαδικασία, γιατί έρχεται η στιγμή πρέπει να πούμε ένα ναι ή ένα όχι. Δεν γίνεται όμως αυτό να γίνεται πάντα αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η πολωνική τότε, η κυπριακή μετά Προεδρία βρήκαν έτσι έναν δρόμο για επικοδομητικό διάλογο με τη συμμετοχή στις άτυπες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναπτύξουμε και να απαιτήσουμε. Ιδάλλως θα πρέπει πάντα να προσφεύγουμε στο ατομικό όπλο. Και επίσης αναφερθήκατε στο χρονοδιάγραμμα του Πρόεδρου Τούσκ. ότι θα έκανε ο πρόεδρος Τούσκ διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Το θέμα είναι ότι η συνθήκη λέει ξεκάθαρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει νομοθετικό ρόλο. Δεν είναι νομοθέτης. Το λέει ρητά η συνθήκη. Δεν μπορούμε να το μετατρέψουμε σε θεσμικό όργανο με αυτόν τον τρόπο. Παίρνει αποφάσεις όσο ισχύει η ομοφωνία. Ιδάλλως πάει από φαστερότατα όργανα και ποιος υπουργό Υπουργείου τολμάει να αντισταθεί σε απόφαση που έχει λάβει ο αρχηγός της κυβέρνησής του στο, στη Συνοδοκορυφή. Μα αυτή η κατάσταση όμως έχει προχωρήσει ε, μέχρι το παράλογο. Έχει φτάσει στο παράλογο αυτή η κατάσταση. Έπρεπε δυνάμει της Λισαβόνας να έχουμε προχωρήσει την περισσότερη, ε, σε περισσότερες ε, εξουσίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το αντίστροφο. Επίσης, φιλόδοξη διαδικασία για έγκαιρη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και νομοθετική βάση μπορεί να υπάρξει εάν η διαδικασία ε, αλλάξει ριζικά προκαταβολικά και όχι με μια πρόταση επιτροπής που μας φέρνει, κατατίθεται το Μάιο και μας φέρνει να περάσουν μερικού μήνες πριν μπορέσουν να δώσουν το τυποθήτο τα όργανα του Συμβουλίου. Πρέπει δηλαδή αμέσως όλα αυτά να προχωρήσουν. Έχουμε τους καθοριστικούς μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο, γίνεται η ψηφοφορία Φεβρουάριο στην ε, Επιτροπή των Προϋπολογισμών, πάει και στο Συμβούλιο του Φεβρουάριο, πάει στον, ε, στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, πάει το Μάιο για έγκριση με μια πολύ συντονισμένη και στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε πολιτικό επίπεδο. Ιδάλω το φιλόδοξο αυτό χρονοδιάγραμμα, το οποίο εμείς το επιδιώκουμε, δεν μπορεί να λειτουργήσει και κύριε Δόκτωρ Μπέγκερ τότε κινδυνεύουμε με ρήξη. Κάνει μια προετοιμασία δηλαδή το τωρινό κοινοβούλιο, έρχεται μετά να ε, συσταθεί, να σχηματιστεί το επόμενο μετά τις εκλογές και μετά ξέρουμε ότι μας έχουν πουλήσει και μας έχουν αγοράσει. Καλύτερα μας έχουν προδώσει και μας έχουν αγοράσει. Άρα λοιπόν καλό είναι να δούμε ποια διαδικασία μας βρίσκει σύμφωνο, σε ποια καταλήγουμε και ποια είναι η βασική συμφωνία στο πλαίσιο της οποίας μπορούμε να εργαστούμε. Η Πασαρέλα, το στάδιο μετάβασης, όντως ε, για την ε, μετάβαση του Συμβουλίου, δηλαδή στην ειδική πλειοψηφία, δεν το θέλησαν δυστυχώς κάποια αρκετά κράτη-μέλη. Αν όμως συνεχίσουμε να ε, το αγνοούμε, αν εμείς τουλάχιστον δεν το θέτουμε, τότε θα αποτύχουμε σε όλα τα θέματα. Πριν από 1,5 χρόνο με τις αλφομπέρες είχαμε τον προϋπολογισμό εδώ στο Κοινοβούλιο. Πολλά θέματα στην έκθεση αυτή, η οποία δεν ζήτησε νέα θεσμικά όργανα, αλλά μίλησε για το Κοινοβούλιο το δικό μας το σώμα, το οποίο είναι αυτό το οποίο είναι αρμόδιο για το ευρώ. Γιατί τα κράτη πλην Βρετανίας και ε, Δανίας έχουν την τάση, αν δεν είναι ήδη στην Ευρωζώνη, να ενταχθούν. Και άρα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ότι ο καθένας έχει συμφέρον να μην επαναληφθεί η κρίση, να προετοιμαστούμε για ενδεχόμενο νέα κρίση, να αναζητήσουμε μία λύση με μία γραμμή στον προπολογισμό, όπως θέλετε πείτε την, για τη σταθεροποίηση του νομίσματος μέσα στην Ευρωζώνη, αλλά ταυτόχρονα μία λύση που δεν θα αποκλείει και τους άλλους εφόσον τους πλήξει κάποια κρίση οικονομική. Τέτοιες λύσεις μπορούμε να τις βρούμε, μπορούμε να τις συμφωνήσουμε και σχετικά γρήγορα, γιατί υπάρχουν τα μέσα και μπορούμε να εξασφαλίσουμε και τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και να καλυφθούμε και εναντί αποφάσεων των Εθνικών Σταγματικών Δικαστηρίων σε σχέση με την εσωτερική ε, ένομη τάξη, ώστε να μην χρειαστεί συνταγματική μεταρρύθμιση στα κράτη αυτά, για να θεωρείς τα κράτη αυτά, πρέπει να είναι τα κράτη, τα κοινοβούλια των κρατών μελών ε, αρμόδια για την απόφαση που αφορά τα έσοδα, αλλά ταυτόχρονα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει τη θέση του μέσα σε αυτό το μηχανισμό, ενδεχομένω σε συνεργασία με έναν αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με του υπουργού των οικονομικών των ε, κρατών τη Ευρωζώνη για, μια ε, διαδικασία σταθεροποίηση σε περίπτωση κρίση του ευρώ. Όταν μπορέσουμε στη Γερμανία να εξασφαλίσουμε μια κυβέρνηση, περιμένω με πολύ μεγάλη αδημονία να δοθεί η ευκαιρία για συζήτηση των προτάσεων του Προέδρου Μακρόν. Ε, ευχαριστώ, κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για το χρονοδιάγραμμα πρώτα. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική ισχύ του Επιτρόπου Έτιγκερ, την εμπειρία της Επιτροπής μας, την στιγμή αυτή κοινωνική και οικονομική, προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία αυτή τη θητεία και αν τα καταφέρουμε καλό θα ήταν. Πολλοί βάζουν το θέμα της νομιμότητας. Λένε ότι αν μιλήσουμε για ένα προπολογισμό πενταετή, το αποκλείσαμε εμείς αυτό, θα ήταν πάντα η προηγούμενη επιτροπή που υποβάλλει πρόταση για την επόμενη επιτροπή. Γιατί οι διαπραγματεύσεις παίρνουν πολύ χρόνο εκτός εάν ελπίζουμε, βάλουμε προθεσμίες και θελήσουμε να πάμε πιο γρήγορα. Η ερώτηση μου είναι, πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιμο στη θητή αυτή να εγκρίνουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεύτερον, γνωρίζοντας τι σημαίνει από πλευράς GNI το, όλα αυτά τα μέσα, τα, καταπεσ... τα κατι καταπιστεύματα, τα διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα. Και εγώ είμαι υπέρ ενός ενιαίου προπολογισμού, αλλά ξέρουμε ότι στις χώρες μέλη έχουν στο μυαλό τους το 1% του GNI ή 1,23% το πολύ. Αν δηλαδή βάλουμε στον προπολογισμό αυτά που είναι εκτό προπολογισμού για να μειώσουμε τον προπολογισμό, ε, καλύτερα να πούμε όχι. Αλλά χρειαζόμαστε τον ενίο χαρακτήρα του προπολογισμού. Να ξέρουμε όμω ότι άπαξ και βάζουμε κάτι μέσα στον προπολογισμό, τότε πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση. Ο δημοκρατικό έλεγχο φυσικά θα ήταν πολύ θετικό αν ήταν όλα μέσα στον προπολογισμό, γιατί θα υπήρχε και περισσότερη διαφάνεια. Ποιο είναι τώρα ο αντίκτυπο, οι συνέπειε, Δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα στον προπολογισμό για να μειώσουμε τον προϋπολογισμό. Ο ενίος χαρακτήρας δεν είναι γι' αυτό το σκοπό. Τώρα, όσον αφορά τον προπολογισμό για την Ευρωζώνη, θα αλλάξουμε όνομα νομίζω. Το να λέμε προπολογισμό τη Ευρωζώνης δεν στέκει με την πρόταση που θα κάνει η Επιτροπή το Δεκέμβριο. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω η Επιτροπή θα κάνει μία πρόταση προκειμένου να είναι ένα backstop για την Τραπεζική Ένωση, τις μεταρρυθμίσεις. Θα μπορούσε να ήταν για την Ευρωζώνη αλλά και για τις χώρες μέλη που θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωζώνη. Άρα η ονομασία δεν ανταποκρίνεται καλά, γιατί δεν περιλαμβάνει όλους τους στόχους. Θα ήθελα και γι' αυτό το τελευταίο το σχόλιο σας παρακαλώ. Πριν να σας δώσω το λόγο κύριε Λένα, ο κύριος δεν πρέχει το λόγο παρακαλώ. Α, θα είμαι λακωνικός γιατί εστερνίζομαι πολλά από τα σχόλια των προλαλισσάντων. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι ε, εκτίμησα ιδιαίτερος αυτό που είπε ο καλεσμένο μας για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ότι είναι μια έννοια δύσκολο να προσδιοριστεί. Πάντως, παρόλα αυτά, η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία είναι μια χρήσιμη έννοια. Χρήσιμη γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα κατά των ευρωσκεπτικιστών. Αρκεί να πούμε ότι το α μέτρο έχει αναφυσβήτητη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα βρείτε να πάσα στιγμή κάποιον τεχνοκράτη να σας το επιβεβαιώσει. Ε, οπότε έχει σημαντικό ρόλο επιχειρηματολογίας για την κατάρρευση του ευρωσκεπτικισμού. Γιατί αν πρέπει να προσδιορίσουμε την προσθέμενη αξία θα έχουμε τέρμονες συζητήσεις. Επίσης, σε αυτή τη φάση θα ήμουν ιδιαίτερα ε, προσεκτικός ε, για τις, ως προς τις μελλοντικές μας αποφάσεις για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί στο μέτρο που τα κράτη-μέλη δεν ξέρουν τι θα γίνει με το Brexit, γιατί και εγώ αν ήμουν αρχηγός κράτους, θα ήθελα πρώτα να δω πόσο θα ε, προσφέρουν οι Βρετανοί για το Brexit πριν εμπλακώ σε τέτοια συζήτηση για τα όρια του προϋπολογισμού. Επίσης, μπαίνουμε σε αχαρτογράφη τα πολιτικά είδατα. Υπάρχει μια πολιτική αβεβαιότητα σε πολλά κράτη-μέλη και αρχίζουν και ανακύπτουν κάποια πολιτικά κινήματα που έχουν σοβαρές επιφυλάξεις για διάφορα πράγματα. Οπότε και το πολιτικό πλαίσιο λήψη αποφάσεων θα επηρεαστεί από τις εξελίξεις που θα λάβουν χώρα μέχρι τη στιγμή της λήψης αποφάσεων. Τρίτον, για τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Εγώ θα ήμουν υπέρ ενό προπολογισμού τη Ευρωζώνη, ε, αν ε, και όπως είπε ο Χωσέ Φερνάντε, θα πρέπει να τον αποκαλέσουμε με διαφορετικό όνομα. Θεωρώ ότι αν ο προπολογισμό τη Ευρωζώνης δεν είναι ο πυρήνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλυθεί σιγά σιγά. Θα εξανεμιστεί. Και το να δώσουμε μια δημοσιονομική ικανότητα στην Ευρωζώνη ίσως έχει ενδιαφέρον για πολλές χώρες ε, και την προσπάθεια ε, περιορισμού της πολιτικής συνοχής. Γιατί λέτε ότι ε, θέλουμε να βοηθήσουμε ε, χώρες για να συνδεθούμε την Ευρωζώνη και θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνοχή στην Ευρωζώνη και να βοηθήσουμε τις χώρες που θέλουν να προσχωρήσουν για να λάβουν επιπλέον ε, κονδύλια για να πραγματοποιήσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για να ενσωματωθούν στην Ευρωζώνη. Ουσιαστικά κάνουμε κάτι θετικό. Δεν στερούμε από κάποιες χώρες ε, το πλεονέκτημα της συνοχής, αλλά προσδιορίζουμε κάτι που τίθεται σε ισχύ και που έχει συγκεκριμένο στόχο τον οποίο συμμερίζονται όλοι. Φανταστείτε ε, σε κάποιες χώρες να πούμε ότι θα μπουν χρήματα στα ταμεία της ε, Ευρωζώνης ενώ θα μειωθούν τα ταμεία συνοχής. Δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσει κανένας αυτό. Θα πρέπει να βρούμε μια συμφωνία που θα έχει θα φέρει πλονεκτήματα και για τις χώρες εν ώψη της μελλοντικής τους ένταξης στην Ευρωζώνη. Τώρα, ως προς τους στόχους του μελλοντικού πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου, δεν θα επισέλθω στο θέμα της αναζήτησης και της οργάνωσης διάρθρωσης της ευελιξίας. Θα βρούμε τρόπο να την επιφέρουμε. Τώρα, ως προς τους πολιτικούς στόχους είμαι πεπισμένο ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε κάποιους πολιτικού πολιτικούς στόχους, όπως ε, τη μετανάστευση. Δεν θα αμβληθούν οι μεταναστευτικές ε, πιέσεις. Το αντίθετο. Ακόμη και αν ε, ελέγξουμε καλύτερα τα τουρκικά και λιβικά σύνορα, δεν θα χαλαρώσουν οι μεταναστευτικές εντάσεις, ούτε θα εκλείψει η τρομοκρατική απειλή. Οπότε όλες αυτές τις προκλήσεις θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη και να μην ξεχάσουμε και το έλλειμμα εμπιστοσύνη των λαϊκών τάξεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι πεπισμένο ότι το μελλοντικό πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο δεν πρόκειται να γίνει όταν έχουμε πανηγυρικά διακηρύξει τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία κοινωνική ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Πώς θα πείσουμε τους πολίτες που προβληματίζονται ε, για το προστεί όλα αυτά που κάνουμε, να κάνουμε κάποιες πανηγυρικές και στο διακηρύξεις και στην πράξη να μην βλέπουν καμία διαφορά. Οπότε, νομίζω ότι οι στόχοι μας είναι σαφής Αλλά προσοχή στο χρονοδιάγραμμα, στους τρόπους εφαρμογής και στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε ως τις πολιτικές μας προτεραιότητες και όχι μόνο ως προς τους μηχανισμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σλένα. Κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου απλώς να αντιδράσω στο θέμα της, ε, του ενίου χαρακτήρα του προπολογισμού. Νομίζω ότι είναι σαφές για την Επιτροπή <clears throat> ότι ο ενίος χαρακτήρας του προπολογισμού είναι πολύτιμος και αν κατά μία περίοδο πολιτής δημοσιονομικού πλαισίου, πλαισίου ε, δεν ε, έχουμε άλλες λύσεις διδικές, για παράδειγμα, αξίζει τον κόπο να διαπραγματευτούμε ένα νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο όπου θα επανέλθει κάποια τάξη σε αυτό τον γαλαξία, όπως τον έχουμε πει, ε, χρηματοδοτικών μέσων. Αυτό είναι μία πτυχή Δηλαδή τι ειδικά μέσα έχουμε στον κανονισμό του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Θέλουμε σε αυτά τα ειδικά μέσα στο μέλλον να προσθέσουμε κι άλλα. Κατά τη γνώμη μου, αυτό έχει να κάνει με την ρυθμιστική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εκτός οροφής και είναι κάτι που μπορεί να κινητοποιηθεί μόνο από τη Δημοσιονομική Αρχή στον ετήσιο προπολογισμό. Άρα να μην θεωρηθεί σαν δορυφόρος, αλλά σαν ένα τακτικό μέσο προπολογισμού. Με την αρχή αυτή, ότι δηλαδή πρέπει να έχουμε όσο γίνεται πιο ενιαίο χαρακτήρα του προπολογισμού, η κατάσταση όσον αφορά το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο απαιτεί πολύ προσοχή. Και θα πάρω το παράδειγμα ανανέωσης παλιότερων δορυφόρων που είχαμε για δεκαετίες, ας πούμε το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τα τελευταία δέκα χρόνια ετοίμασαν τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο να μπορεί να ενσωματωθεί στον τακτικό προπολογισμό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί για αυτό το σκοπό και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να ενσωματώσουμε το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο στο κυρίω σώμα του προπολογισμού. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι κάτω από αυτές τις ειδικέ συνθήκες πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το πώς θα το κάνουμε, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η ενσωμάτωση του Αναπτυξιακού Ταμείου δεν θα μειώσει τις δυνατότητες για αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί αυτό τότε θα αντέβαινε στις πολιτικές προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι εύκολη η δουλειά και για κάποιο λόγο που ακούσαμε στην προηγούμενη συζήτηση που υπογράμμισε η κυρία Ρούμπιο ότι δηλαδή η οροφή για τους ίδιους πόρους θα επηρεαστεί από την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και η οροφή αυτή ιδίων πόρων, ίσως ο κύριος Μπέκερ θα μπορούσε να ενημερώσει την παρουσίασή του, γιατί από το 2016 ισχύει ένα νέο λογιστικό σύστημα και είναι 1,20% η οροφή του Ευρωπαϊκού GNI. Αυτή η οροφή λοιπόν σε απόλυτα ποσά θα μειωθεί σημαντικά αν υπολογιστεί με βάση τις 27 χώρες και όχι τις 28. Και αυτό θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τον ετήσιο προπολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υποχρεώσεις που πρέπει να φέρουμε σε πέρας με την ίδια οροφή. Και εκεί είναι που μαζί πρέπει να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε η ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου να γίνει χωρίς να επηρεαστούν τα κονδύλια για την αναπτυξιακή πολιτική και να είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε στα κράτη-μέλη ότι μπορεί να χρειαστεί να αυξηθεί το όριο ιδίων ε, πόρων ακριβώς επειδή ενσωματώνουμε διάφορα μέσα τα οποία μέχρι τώρα λειτουργούσαν ως δορυφόροι και τώρα τα ενσωματώνουμε μέσα στο κυρίω σώμα του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Δύσκολο να εξηγήσουμε το εγχείρημα, αλλά γι' αυτό το σκοπό θα έπρεπε να αυξηθούν οι ήδη Και μία παρατήρηση για το χρονοδιάγραμμα τέλος. Ο Επίτροπός μου, ο Επίτροπος Σίτιγκερ, έχει πει ότι θέλει διακόστο το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να προχωρήσουν γρήγορα σε διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν αυτές γρήγορα με επιτυχή κατάληξη κυρίως για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τον ε, επόμενο προπολογισμό. Ευχαριστώ. Ähm, Ευχαριστώ. Έφτασε και ο κύριος Πόνς. Και είμαι αποφασισμένος να του δώσω το λόγο στις 5. Μας μένουν 15 λεπτά λοιπόν. Γι' αυτό, εάν τυχόν δεν έχετε κάτι άλλο, ή να ξεκινήσουμε με τον δόκτωρα Μπέκερ. Σχόλια, συνοψίζετε, απαντάτε. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και για τα σχόλιά σας. Θα είμαι λακωνικός. Καταρχήν ως προς τη θέμενη αξία. Όπως είπα, είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε αυτή την έννοια. Η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε επιμακρό να, να προσδιορίσει αυτή την αρχή της θέμενη αξία και το 2009-2010 μάλιστα δημοσίευσε ε, μετά από χρονοβόρες συζητήσει. Το 2011 δημοσίευσε το έγγραφό της και το συμπέρασμά της ήταν ότι μπορεί κανείς να βρει την προστιθέμενη αξία εξετάζοντα τα ποσά του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, αυτό το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων δηλαδή είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτό ήταν το πολιτικό συμπέρασμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τι εστί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ως προς το χρονοδιάγραμμα σας ε, παρουσίασα συγκριτικά τα χρονοδιαγράμματα από τις εμπειρίες των προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Αν προβάλλετε τα παλιά χρονοδιαγράμματα στην παρούσα κατάσταση, θα καταλήξουμε στις αρχές του 2020 για το πέρας των διαπραγματεύσεων. Για να είμαστε ρεαλιστές, ε, ε, πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να διαπραγματεύεται για συγκεκριμένα νούμερα, για ποσά, για αριθμούς, γιατί τα κράτη-μέλη δεν είναι σίγουρο ότι θα καταλήξουν συμβαστική λύση μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους. και τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης ή τη δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης, είναι ακόμη ασαφές πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτή η δημοσιονομική ικανότητα ή αυτός ο προϋπολογισμός της Ευρωζώνης, ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες του, αν θα είναι μικρή σχετικά ικανότητα και θα αφορά τη χρηματοδότηση μόνο εθνικών μεταρρυθμιστικών αναγκών ή θα είναι τεράστιος ο προπολογισμό 1-2-3% του ΑΕ, του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ευρωζώνης. Ε, ή θα προσπαθήσει να καλύψει κυκλικές ανάγκες, ε, να χρηματοδοτήσει προγράμματα, να σταθεροποιήσει τη νευροζώνη και να ασκήσει πραγματική πολιτική στην Ευρωζώνη. Είναι ανοιχτό ακόμη αυτό το θέμα, τι θα εξυπηρετεί ένας τέτοιος προϋπολογισμός. Πάντως ένας μεγάλος ε, προϋπολογισμός της Ευρωζώνης που ήταν η ιδέα του Παρισιού αρχικά προϋποθέτει ένα προϋπολογισμό θα περιλαμβάνει κάθε χρόνο πάνω από 230 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή θα είναι σχεδόν διπλάσιος από τον τρέχοντα προϋπολογισμό για τους 28. Ε, ε, και θα χρηματοδοτεί υποδομές, ε, καινοτομία, ανάπτυξη. Τώρα, σε σχέση με τις ισχύουσες προτεραιότητες για τις δαπάνες, έχουμε τα διαρθρωτικά ταμεία με τις ίδιες αρμοδιότητες. Οπότε, ένας νέος τέτοιος προϋπολογισμός προϋποθέτει συμφωνία ως προς την περιπλοκότητα και την αδιαφάνεια και θα επιτείνει τον κατακαιρματισμό. και θα καταστήσει σαφές ποιος είναι πραγματικό πυρήνας για τη μομηχανή της Ευρωπαϊκής Χάραξης Πολιτικών. Ευχαριστώ, Γιάννου Ευχαριστώ πολύ. Επανέρχομαι στο αρχικό σας σχόλιο ότι καλή είναι η προσθέμενη αξία, αλλά δεν είναι στόχος. Είναι ένα μέσον για την επίτευξη του στόχου. Εάν πούμε ότι στόχος μας είναι να δουλεύουμε καλύτερα, δεν θα, μείνουμε και πολύ, θα ήμασταν και πολύ φιλόδοξοι. Επομένω, πρέπει να έχουμε κάτι καλύτερο, περισσότερη αξία. Μέχρι τώρα δηλαδή κάναμε κάτι το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα αξιόλογο. Α το κάνουμε καλύτερα. Α είμαστε φιλόδοξοι. Η πολιτική τη Ευρώπη του ή άλλω είναι να πείθει τους ε, λαϊκιστές ότι δεν πρέπει να είναι λαϊκιστές. Κοιτάξτε, είμαστε πολιτικό σώμα εδώ. Και αυτή είναι η δουλειά μας. Να αποφασίζουμε τι θέλουμε. Θέλουμε κοινότητα ή θέλουμε διακυβερνητική. Αυτό είναι το ερώτημα. Αν είναι καθαρά διακυβερνητική η λύση, ευρωπαϊκό προπολογισμό. Δεν χρειάζεται. Κανένα από αυτά σενάρια. Ούτε καν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται. Ναι, αυτό είπα και στον Τσέχο Πρωθυπουργό που είπε ότι δεν χρειάζεται Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, πρόεδρο της Δημοκρατία, μάλλον, που είπε ότι θέλουμε... δεν χρειάζεται Κοινοβούλιο. Επομένω, το θέμα δεν είναι τα νούμερα, αλλά το μελλοντικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κάποια μέσα για να εξυπηρετήσουμε το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουμε για το οποίο αγωνιζόμαστε. Εκεί λοιπόν πρέπει να διαρωτηθούμε. Τι είναι αυτό που είναι πιο ευέλικτο, στο οποίο μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις, ποια είναι η δυναμική του, σε τι αναλογία στέκεται το κάθε του σκέλος προς τα υπόλοιπα. Και ευχαριστώ που μας λέτε τι είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωζώνης. Ό,τι όνομα και να του δώσουμε. Όπου και να τον κρύψουμε πίσω από ωραίες εκφράσεις. Ο προπολογισμό της Ευρωζώνης είναι. Είναι τα ίδια μέσα για το ευρώ, μέσα στον προπολογισμό, αλλά για ένα μέρος των χωρών. Και ας το πούμε, ας πούμε την αλήθεια, ο προπολογισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αφορά κάποιους και κάποια πράγματα, κάποιες πολιτικές, ενώ ο προπολογισμό Ευρωζώνης θα αφορά κάποιους άλλους και, τομεί και ε, τομείς του εις Ευρωζώνης. Αν πρόκειται για χώρες εκτός της Ευρωζώνης θα έχουμε τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεξής. Αλλιώ θα είναι τα ταμεία, θα τα λέμε, θα το ονομάζουμε αλλιώ κτλ. Αυτά συνοψίζοντα. Επομένω, η συζήτηση για το πουδουπού δεν είναι για το χρήμα. Είναι η συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το πώς θέλουμε να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς προσπαθούμε να εκφράσουμε σε δημοσιονομικούς όρους πολιτική σκέψη. Αυτά. Γκάιερ. Ευχαριστώ την κυρία Ρούμπιο, τον δόκτωρα Μπέκερ, τον κύριο Λενά, την νομική μας υπηρεσία. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. και ενημερωτικά. Προχωρήσαμε, είμαστε και λίγο πιο μπροστά από το χρόνο μας, έχουμε 5-6 λεπτά παραπάνω. Κύριε Πόνς, μια έξετε εδώ, ας περάσουμε στο δικό σας θέμα αναπτυξιακό πρόγραμμα για πρόγραμμα ανάπτυξη μάλλον της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας που είναι συνδεδεμένη Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης σε θέματα άμυνας. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για όλους μας, γιατί στόχος του είναι να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της Ευρώπης. Η πρωτοπορία η τεχνολογική έχει κέρια σημασία και αυτό θα πρέπει να ισχύει και για μας. Και επίσης θα πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία, να δώσει ανάπτυξη για τη συνεργασία για να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα και, τη, και να βελτιστοποιήσει και την ποιότητα των αμυντικών δαπανών. Επίσης θα πρέπει να συνεργάζονται και οι άνοπλες δυνάμεις μας μεταξύ των κρατών μελών και ευτυχώ έχουμε συμφωνήσει όπως το μόνιμο τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία που στις 13 Νοεμβρίου την υπέγραψαν 23 από τι 28 χώρε μέλη. Η μέχρι στιγμής έλλειψη συνεργασίας μας στοιχίζει 25 με 100 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και αυτό γιατί περίπου 80% των δημοσίων έργων για την άμυνα δίνονται σε εθνικό επίπεδο των κρατικών προμηθειών για την άμυνα, κάτι που δημιουργεί περιτές επικαλύψεις στις άμυνες μας. Το πρόγραμμα αυτό εδράζεται κυρίως και επικεντρώνεται στο σχεδιασμό προϊόντων και αναλυτικών για τεχνολογίες άμυνας, για κοινέ τεχνολογικές προδιαγραφές, δημιουργία πρωτοτύπων και δοκιμών, και εκπόνηση κάποιων μελετών. Επίσης, ε, έχουμε, θα πρέπει να έχουμε συνεργασία τουλάχιστον τριών επιχειρήσεων με ε, έδρα τουλάχιστον σε δύο χώρες μέλη. Για τη χρηματοδότηση προβλέπονται 500 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2019-2020. Είναι λογικός κατά τη γνώμη μου αυτός ο προτινόμενος προϋπολογισμός. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο ποσό θα πρέπει να προέλθει από τα περιθώρια του δημοσιονομικού πλαισίου, γιατί νέες πρωτοβουλίες που θα είναι υποφελείς για όλους δεν πρέπει να χρηματοδοτεί εις βάρος άλλων ε, προγραμμάτων ή πολιτικών που δεν έχουν καμία σχέση με τις καινούργιες προτεραιότητες. Και να μην ξεχνούμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι κινητήριος δύναμη της οικονομίας μας. Και τουλάχιστον μία κατηγορία σχεδίων θα πρέπει να αφιερώνεται ιδιαίτερως σε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης να εξασφαλιστεί το 20% τουλάχιστον 100 του συνολικού προϋπολογισμού να αφιερωθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για να διευκολυθεί η εφαρμογή του προγράμματος και να εγγυηθούμε την επιτυχία του, ζητούμε με την γνωμοδότηση να δώσουμε την, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, την, ε, την εξουσία να υιοθετήσει τις εξουσιοδότηση πράξης για το πρόγραμμα εργασιών. 7 Δεκεμβρίου λίγη ιδεωρία για την υποβολή τροπολογιών στις 3 το απόγευμα. Αυτά και είμαι ανοιχτό στις προτάσεις ε, και τα σχόλια των συναδέλφων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Βονσέλης Πόνς. Μόνο εγώ έχω ζητήσει το λόγο. Α, ο κύριος Κολόν. Ναι, ναι, ναι. Σας, σας είδα, σας είδα. Αυτό ήθελα να πω. Κάποιον άλλον δεν είδα. Κύριος Δουρανού. Δεν θέλω επί της ουσίας να τοποθετηθώ, όχι ως προεδρεύων αυτή τη στιγμή, αλλά ως μέλος της Επιτροπής. Πρόκειται για τη θέση της σοσιαλδημοκρατικής αντιπροσωπείας από τη Γερμανία των σοσιαλδημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή δεν έχω συστήσει το θέμα με τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ούτε καν είμαι σκιώδης συγητής. Απλώς εκφράζω το S5 της Γερμανίας την αντιπροσωπεία του εδώ, που έχει κάνει μια συζήτηση για το θέμα αυτό και το πρόγραμμα. Πρώτον, η νομοθετική βάση είναι προβληματική εδώ, η νομική βάση, διότι υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της νομικής βάσης που έχει επιλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στηρίζεται στο ότι πρόκειται για πολιτική ε, βιομηχανική και άλλου άρθρου της συνθήκης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει ρητά τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει δραστηριότητες στον τομέα, που απαγορεύει συγγνώμη, ρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση την αναπτύξη δραστηριότητες στον τομέα των εξοπλισμών. Οπότε το ορίζον 2020 μάλλον δεν πρέπει να μπει σε, αυτό, σε αυτή τη συζήτηση. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι καλή επιλογή τη νομική βάση για το πρόγραμμα. Και σας καλώ να το σκεφτείτε όλοι. Δεύτερον, αξιολόγηση είναι η επόμενη ερώτηση. Ο καθένας μπορεί να καταλήξει διαφορετικά συμπεράσματα. Πιστεύω ότι το δυναμικό εξοικονόμηση που μας προτείνεται ως προοπτική είναι θεωρητικό. Ήμουν βουλευτή άλλου. Ήμουν βοηθό άλλου βουλευτή όταν ξεκίνησε η ενιαία αγορά και υπήρξε μια ευρωπαϊκή οδηγία για το χώρο των κατασκευών όπου ήταν απόλυτο σαφές ότι ο κατασκευαστικός κλάδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να ενοποιήσει κάποιες δραστηριότητες με ένα τεράστιο δυναμικό για εξοικονόμηση πόρων, μείωση δαπανών. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ούτε πρίζες δεν έχουμε ίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλοι τρέχουμε με έναν αντάπτορα στην ε, τσάντα και μας πιάνει πανικός αν τον έχουμε ξεχάσει και φτάσουμε το βράδυ στο ξενοδοχείο και δεν έχουμε τρόπο να φορτίσουμε. Μήνες και συζητήσεις και ειδική ε, διφασικός, τριφασικό, ε, διφασική, τριφασική πρίζα ε, ε, ηλεκτρικού πέρασαν και σβήστηκαν με μια πολύ λακωνική και χαρακτηριστική φράση ότι δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να εναρμονίσει τα πάντα μέχρι και το καπάκι της τουαλέτας. Έτσι λοιπόν, μπορεί να προσπαθεί ο καθένας να προστατεύσει τον τομέα του και φαντάζομαι ότι αυτό συμβαίνει τώρα με, την, ε, ε, με τον κλάδο της βιομηχανίας ε, εξοπλισμών και άμυνας και αυτό σημαίνει ότι η κάθε κυβέρνηση θα προσπαθήσει να σε κάθε είδους κίνδυνο ανταγωνισμού εις βάρος της οικίας της βιομηχανίας όπλων. Αυτό είναι λογικό. Πρόκειται για δημόσιο κλάδο, πρόκειται για κράτος. Τώρα, τώρα προχωρήσει κάπως διαφορετικά η ιστορία θα με εξέπλητε πολύ. Τρεις εταιρείε από δύο κράτη-μέλη τουλάχιστον δείχνουν να ενδιαφέρονται και να δίνουν ενδείξεις προς την κατεύθυνση αυτή, διότι εάν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, αυτή η προοπτική, δεν θα είχε καν λόγο να δραστηριοποιηθεί στον τομέα αυτό των συνδικών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης, και χαίρομαι ιδιαίτερος ε, κυρία Κονσάλες Πόνς για τη θέση σας στο σημείο αυτό, το θέμα της χρηματοδότησης. Γιατί κατατρόμαξα όταν η Επιτροπή, όχι εδώ σε αυτή, αλλά στη δική μας Επιτροπή, έκανε πρόταση για χρηματοδότηση και όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει για τα ανεπαρκή περιθώρια του πουλέτου του νοσονομικού πλαισίου, για ανελεκτικέ πηγές χρηματοδότησης, ε, παίρνουν ακόμη πιο εναργείς διαστάσεις εάν έρθει και το θέμα του, ε, της χρηματοδότησης του τομέα της άμυνας και των εξοπλισμών εδώ μέσα. Γι' αυτό λοιπόν και εκ μέρου επαναλαμβάνω τις αντιπροσωπία μου και όχι της ομάδας μου σας δηλώνω ότι το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσαμε να το δεχθούμε μόνο εάν προκύψουν νέες φρέσκες νοπές πηγές χρηματοδότησης για το τομέα αυτό και ο συνάδελφος έχει το λόγο. Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή. Και συνεχίζω ακριβώς τη δική σας γραμμή και τις επιφυλάξεις κύριε Γκάιερ είναι με το συμπάθειο που θα το πω έτσι, πολύ απρόσεκτη η προετοιμασία αυτής της ε, υπόθεσης. Δεν το έχετε σκεφτεί καλά. Μπορεί να ακούγονται πολύ ωραία όλα αυτά. Μπορεί ο, το δυναμικό παραγωγής των ε, ε, στρατιωτικών δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να πούμε ότι θα ενοποιηθεί. Αλλά εδώ δεν μιλούμε για ψίχουλα, μιλάμε για δισεκατομμύρια σε ευρώ έχει κάτσει κανείς να σκεφτεί σε όρους οικονομικούς με βάση την απόδοση και τις τιμές και τις οικονομικές κλίμακες όλα αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βελτιώσουμε κάτι που ήδη είναι αρκετά καλό. Βεβαίως και μπορούμε. Αλλά ταυτόχρονα η προσέγγιση είναι προσέγγιση που μας οδηγεί σε εσφαλμένα αποτελέσματα αν θεωρούμε ότι πρέπει να χτίσουμε ένα κλάστερ, έναν θύλακα, γιατί αυτό δεν θα μας εξασφαλίσει περισσότερο ανταγωνισμό ή περισσότερη προσθέμενη αξία, αλλά μόνο, προσθε... μόνο περισσότερη γραφειοκρατία. Άλλο να θέλει κανείς και ο θελός να πει ότι να συνενώνω τις δυνάμεις μου και το κάθε κράτος αποφασίζει μόνο του αν θέλει να συμμετάσχει σε αυτή τη συνένωση δυνάμεων. Εδώ έχουμε περισσότερα οπλικά συστήματα ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως κράτη Ευρωπαϊκής Ένωσης από ότι το ΝΑΤΟ ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αλλά θα πρέπει και ταυτόχρονα να δούμε εάν είναι διατεθειμένα τα κράτη-μέλη να περάσουν στην εφαρμογή ενός ενιαίου οπλικού συστήματος, ενός μοναδικού οπλικού συστήματος. Γιατί αν μείνουν έστω και δύο διαφορετικά οπλικά συστήματα δεν λειτουργεί το σύστημα. Άρα πρέπει να θέσουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων και να κοιτάξουμε τι ακριβώς είναι διατεθειμένα τα κράτη να ενοποιήσουν. Γιατί μόνο τότε και μόνο αυτό μπορεί να ενοποιηθεί. Αυτό όμως πρέπει να ξεκινήσει από τα κράτη-μέλη τα ίδια. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πλαίσιο μόνο πρέπει και μπορούμε να εγκαθιδρύσουμε που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να έχουν μια πιο αποτελεσματική και γρήγορη ε, δυνατότητα προμηθειών ουσιαστικά. Γιατί από την άλλη πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ταυτόχρονα μπορεί να χαθούν δισεκατομμυρίων αξίας συμβάσεις προμηθειών. Δεν μπορούμε να δεχθούμε τέτοιου είδους οικονομικές απώλειες. Να λέμε ότι πρέπει να αγοράζουμε πιο αποτελεσματικό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα να μην μπορούμε να πολλούμε με τους ίδιους όγκους από την οπλική μας βιομηχανία, δηλαδή για να τη στηρίξουμε να πρέπει να πληρώνουμε επιδοτήσεις. Δεν είναι απλά τα πράγματα όπως τα παρουσιάζετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι είμαστε εδώ στην καρδιά του προβλήματος. Πρόκειται για τεχνικά ζητήματα, δημοσιονομικά, βέβαια. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε σε αυτά για την άμυνα, δηλαδή στην Ευρώπη. Υπάρχει απειλή, το γνωρίζουμε. Οι Αμερικανοί αποδεσμεύτηκαν. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ασχοληθεί με τη δικιά της ασφάλεια και προστασία. Οπότε πολύ με ενδιαφέρουν όλα αυτά που γίνονται γύρω από την ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να έχει περισσότερη συνεργασία μεταξύ της στον τομέα της άμυνας. Έχω δουλέψει για την έρευνα, τώρα μιλάμε για την βιομηχανία, για την παραγωγή δηλαδή εξοπλισμού. Δεν πρέπει απ' την άλλη να ε, τα κάνουμε όλα κουβάρι και να πετάμε το μωρό με τα νερά του μπάνιου όπως λέμε. Πρέπει το θέμα της ε, άμυνας να το δούμε από μόνο του. Δεν είναι απλά. Αν ήταν απλά δεν θα τα συζητούσαμε τώρα, θα την είχαμε ήδη βρει τη λύση. Πάντως, μία από τις κύριες ανησυχίες είναι η οικονομική. Και τα χρήματα για τα οποία μιλάμε δεν φτάνουν σε σχέση με τις ανάγκες που εκφράζονται. Θα έπρεπε λοιπόν πολύ γρήγορα οι χώρες μέλη να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει επιτέλους να δώσουν τα αναγκαία χρήματα για να στηρίξουν αυτή την ευρωπαϊκή άμυνα. Είναι ένα πρώτο βήμα. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες, τις τεχνικές, νομικές και οικονομικές. Αλλά πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Η κυρία Αγαπητοί συνάδελφοι, τρέφω κάθε κατανόηση στο ότι λέμε πως είναι προώρο να συστήσουμε μηχανισμούς ε, πριν να υπάρχει μια ουσιαστική εικόνα, πριν έχουν προσδιορίσει τα κράτη-μέλη και όλα αυτά. Αλλά είναι δυνατόν όλα αυτά να σημαίνουν ότι μένουμε μετακίνητοι και δεν αλλάζουμε τίποτα. Όχι. Πρέπει να μας οδηγεί στην αναζήτηση μηχανισμών, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, και όταν υπάρχει και επειδή υπάρχει ενισχυωμένη απειλή και γιατί αλλάζει το πολιτικό θεματολόγιο και γιατί αφενός μεν από αυτά προκύπτει ότι θα χρειαστεί και περισσότερα να παράγουμε και περισσότερα να αναπτύσσουμε από κοινό και άρα θα πρέπει να σκεφτούμε πόσο μπορούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και επιπροσθέτως τι άλλο χρειάζεται και αυτό που χρειάζεται αφού το βρούμε να το χρηματοδοτήσουμε κι άλλο και επίσης και από το ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και από τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η προσέγγιση που έχει επιλέξει ο συνάδελφος Κονσάλες Πόνς, μια πολύ καλή και σωστή προσέγγιση που λέει να ξεκινήσουμε. Δεν είναι το τελευταίο βήμα αυτό που μας περιγράφει, αλλά το πρώτο βήμα. Και να κοιτάξουμε, να εξετάσουμε και να δώσουμε απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Πρώτο βήμα λοιπόν, θα ακολουθήσουν άλλα βήματα, πρέπει να τα συζητήσουμε αφού το αναλύσουμε πρώτα. Ευχαριστώ πολύ και καλό την Επιτροπή να τοποθετεί. Θη, αν θέλει κανείς, παρακαλώ εσείς. Thank you, Mr. Geyer. Ευχαριστώ κύριε Γκάιερ και ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που παρακολουθήσαμε. Ε, ως εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμών θα επικεντρωθώ στα σχόλιά μου στα χρηματοδοτικά θέματα. Με αυτό ασχολούμαι και αυτό απασχολεί και φυσικά τα μέλη της Επιτροπής σας. Θυμάμαι πολύ έντονα ότι τον Ιούλιο σας παρουσίασε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, εδώ στην Επιτροπή σας. Σας παρουσίασε λοιπόν την πρόταση για χρηματοδότηση των 500 εκατομμυρίων κατά 75% με πολλές μεταβάσεις από το Α1 τομέα και 25% από τα περιθώρια που δεν έχουν αξιοποιηθεί από τα χρησιμοποιητά κονδύλια. Και είναι σαφές ότι δεν έγινε πολύ ενθουσιοδός ε, δεκτή πρόταση από την Επιτροπή σας. Θυμάμαι την έντονη αντίδραση του κ. Φερνάντες αλλά και πολλών άλλων κατά της πρότασης. Οπότε είναι σαφές και το μήνυμα ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο θα επιδιώξει συμβασμό που προϋποθέτει πολύ λιγότερες μεταφορές κονδυλίων από επιμέρους δημοσιονομικές γραμμές. Αλλά μην ξεχνάτε ότι και από το Συμβούλιο ε, η θέση φαίνεται να γίνεται όλο και πιο άκαμπτη. Και φαίνεται ότι η πρόθεση του Συμβουλίου στην γενική προσέγγιση τουλάχιστον που προετοιμάζει είναι 100% ανακατανομή των κονδυλίων. Φυσικά δεν μπορώ να προεξοφλήσω την ε, οριστική θέση του Συμβουλίου. Αλλά μέχρι στιγμής αυτή είναι η κρατούσα άποψη στο Συμβούλιο. Υπέρ 100% ανακατανομή των κονδυλίων. Κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την θέση του Συμβουλίου σε προηγούμενη φάση των διαπραγματεύσεων για το ΕΦΣΙ εκεί. Ε, το Συμβούλιο αρχικά είχε δεχτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να κατανομή ε, της τάξης του 75%. Οπότε στο μέτρο που προχωρούν οι διαπραγματεύσεις το Συμβούλιο σκληραίνει τη θέση του. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτή τη φάση μπορούμε μόνο να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι διαπραγματεύσεις για την χρηματοδότηση πρόσθετες αυτής θα είναι πολύ επίπονες και ελπίζω να υποβληθούν συμβαστικές προτάσεις ε, ε, για να βοηθήσουμε και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξουν και εγκαίρως σε συμφωνία για την πολύ σημαντική αυτή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης παρούσα. Από ό,τι ξέρω θέλετε να λάβετε το λόγο. DG Grow. Euh, Ευχαριστώ. Μια παρατήρηση, ένα σχόλιο. Και κάτι σημαντικό που έχει με την, να κάνει με την νομική βάση. Πράγματι, πρέπει να γίνει η διακρισή ανάμεσα στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 173, που αποτελεί βάση για την πρόταση αυτή, και τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η δεύτερη απαγορεύει τη χρήση του κοινοτικού προπολογισμού για την συγχρηματοδότηση δράσεων στον τομέα της άμυνας. Και γι' αυτό αυτό το πρόγραμμα δεν βασίζεται στη συνθήκη της ε, Ένωσης αλλά στη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 173 που έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας. Στόχος του προγράμματος δεν είναι η χρηματοδότηση της άμυνας αλλά η βιομηχανία και μόνο στα στάδια ανάπτυξης μέχρι το πρωτότυπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει να πάμε πιο πέρα ούτε προτείνει τη χρηματοδότηση της απόκτησης ικανοτήτων, γιατί αυτό είναι θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας των χωρών μελών. Οπότε πιστεύουμε ότι αυτά είναι απόλυτα συμβατά με τη συνθήκη. Τώρα είναι αλήθεια ότι το πρόγραμμα Horizon 2020 δεν επιτρέπει τη χρηματοδότηση ε, αμυντικών βιομηχανιών. Γι' αυτό και δεν βασιζόμαστε στο Horizon 2020, πήραμε άλλη γραμμή ανεξάρτητη. Είμαστε εντελώς εκτός του προγράμματος ε, Ορίζοντας 2020, ξέροντας ότι υπάρχει ο κανονισμός του Horizon 2020 που αποκλεί τη χρηματοδότηση άμυνας. Η συνθήκη όμως δεν εμποδίζει τη χρηματοδότηση της έρευνας ε, για την άμυνα. Συνεπώς με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, βέβαια εφόσον πρόκειται μόνο για την ανάπτυξη και σταματήσουμε μετά το στάδιο ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις. Ο εισηγητής παρακαλώ, κύριε Κονσάλης Πόνς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ όλους για αυτή τη συζήτηση που είχαμε που είναι μόνο η πρώτη, έτσι. Θα ακολουθήσουν κι άλλες, δίχως άλλο, που θα είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσες. Περιμένω τις τροπολογίες όλων των συναδέρφων και τα σχόλιά σας, ώστε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που να μπορέσει να εγκρίνει η Επιτροπή μας. Όμως, υπάρχουν τέσσερα πράγματα που θα ήθελα να διευκρινίσω. Πρώτον, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα έγγραφο για την ευρωπαϊκή άμυνα. Δεν συζητάμε το κατά πόσο η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να τίνει ε, προς μια ευρωπαϊκή πολιτική άμυνα ή όχι. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση προεπολογισμού σχετικά με την πολιτική η οποία αποφασίζεται σε άλλη επιτροπή. Συνεπώς δεν είμαστε εμείς που θα συζητήσουμε για το κατά πόσο πρέπει ή όχι να ενισχυθεί η αμυντική ευρωπαϊκή βιομηχανία. Μας ε, ζητούν να αποφανθούμε ως Επιτροπή Προϋπολογισμών για ένα θέμα που συζητάει άλλη Επιτροπή που είναι αρμόδια για αυτό το ζήτημα. Δεύτερον, θα ήθελα όλοι να καταλάβουν ότι εδώ δεν μιλάμε για αγορά υλικού, μιλάμε για έρευνα. Δεν λέμε να αγοράσουμε υλικό μαζί όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις άμυνας θα μπορούν να ερευνούν από κοινού μειώνοντας το κόστος των χωρών μελών που συμμετέχουν σε αυτή την έρευνα. Τρίτον, από δημοσιονομική άποψη, είναι προφανές ότι μια από κοινού έρευνα οδηγεί σε εξοικονόμηση πόρων. Γιατί σήμερα δαπανάμε στην έρευνα για την ε, άμυνα 26-27 φορές, ο καθένας δηλαδή, η κάθε χώρα χωριστά. Δεν είναι αυτό εξοικονόμηση πόρων. Φανταστείτε πόσο θα κόστιζε ο στρατός των Πολιτειών αν η έρευνα στην άμυνα δεν ήταν ομοσπονδιακό ζήτημα, αλλά ζήτημα της κάθε πολιτείας χωριστά. Οπότε, αν είχαν ένα μοντέλο τάγκ, ας πούμε, είχαν 51. Αυτό όμως γίνεται στην Ευρώπη. Δαπανούμε περισσότερα από τη Ρωσία στην ε, έρευνα και στην τεχνολογία για την αμυντική μας βιομηχανία η οποία έτσι καλώ βρίσκεται πολύ πιο πίσω από τη ρωσική. Και τελειώνω και με μία σκέψη προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακολουθώντας την ίδια γραμμή σκέψης που ανέφερε και ο Πρόεδρός μας πριν. Εάν εδώ μιλάμε για μια κοινή πολιτική έρευνας στον τομέα της άμυνας, αυτό γίνεται για να εξοικονομήσουμε χρήματα. Η εξοικονόμηση αυτή δεν γίνεται από τον προπολογισμό τον ευρωπαϊκό, αλλά τον προπολογισμό των χωρών μελών. Οπότε δεν έχει νόημα συγχρόνως να λέμε ότι πρέπει από κοινού να ερευνήσουμε στον τομέα της άμυνας για να εξοικονομήσουμε χρήματα από τους προϋπολογισμούς των χωρών μελών και οι πόροι για την κοινή αυτή έρευνα να βγαίνουν από τον κοινοτικό προπολογισμό. Μα αν η εξοικονόμηση θα γίνει στους εθνικούς προπολογισμού τότε να είναι οι εθνικοί προπολογισμοί οι οποίοι θα συνεισφέρουν με περισσότερου πόρου και όχι να αφαιρέσουμε κονδύλια από τον κοινοτικό προπολογισμό. Εφόσον θα εξυπηρετηθούν οι εθνικοί προπολογισμοί, αυτοί να χρηματοδοτήσουν και την αποκοινού έρευνα. Από εκεί και πέρα περιμένω τις δικές σας σκέψεις και σχόλια και προσβλέπω σε μια επόμενη συζήτηση σε βάθος γιατί το θέμα απαιτεί τέτοιου είδου συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κοντσάλης Τα καταφέραμε και πιο νωρί μάλιστα είμαστε έτοιμοι. Πεντέμιση περιμένουν συνάδελφοι να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Επομένω, φαντάζομαι δεν θα έρθουν πιο νωρί. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω αυτά τα 12 λεπτά που μα μένουν να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να είμαστε έτοιμοι 5 και 30 να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Για να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ξέρετε ότι για την ψηφοφορία χρειαζόμαστε τις κάρτες μας. Θα τις έχετε φαντάζομαι όλοι πρόχειρες. Υπάρχει κανείς που να έχει ξεχάσει την κάρτα του να μας κάνει να μας ενημερώσει ώστε να το κοιτάμε όταν σηκώνει το χέρι αναλόγως. Καλά, λοιπόν, μια δοκιμαστική ψηφοφορία παρακαλώ. ας πούμε ερώτημα. Ε, έχω μέχρι στιγμής ε, διαχειριστεί την ε, Προεδρία της Συνεδρίας κατά εξαίρετο τρόπο. Παρακαλώ ψηφίστε υπέρ. Άντε ας ξεκινήσουμε. Δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Αυτό πρέπει να πω. Ωραία. Ψηφίσατε όλοι. Έτσι βλέπω. Πέρα της ψηφοφορίας. είναι κατά, εννέα απέχουν από ό,τι βλέπω, 17 συμφωνούν. Τι μου, εξιδίων τα βέλη. Ψηφίζουμε λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι. Δεν περισσεύει κανένα από τις ε, ομάδες, ε, από, τις, ε, από τους συναδέλφους που ψηφίζουν και ξεκινώ όχι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να επισημάνω ότι έχουμε πολλές ψηφοφορίες που έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής. Τη Παρασκευής της νύχτας που συζητήσαμε και σήμερα το πρωί. Τι στάση θα τηρήσουμε. Πολιτική τοποθέτηση πρώτα σε σχέση με την ε, συνδιαλλαγή γιατί το Κοινοβούλιο είχε πει ότι τον διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 6 για το 2017 θα τον ενέκρινε εφόσον καταλήγαμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα για τη συνδιαλλαγή, όπως και έγινε. Τη δική μου έκθεση λοιπόν ψηφίζουμε πρώτα. Τροποποιητικός Προπολογισμό υπαριθμών 6. Διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 6. ε, τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ με μια ψήφο υπέρ. Απερίφθη 2 υπέρ. Κατά. Δύο ψήφοι υπέρ. Απερίφθη. 3 υπέρ. Κατά. Απερίφθη 4 υπέρ. 5 κατά περισσότεροι εποχές απερίφθη στο σύνολο ονομαστική ψηφοφορία άρχεται Entschuldigung, Entschuldigung, mein Fehler, ich werde... Όχι, δικό μου το λάθος. Ε, πρέπει πρώτα να πω ότι υπάρχουν δύο τεχνικές προσαρμογές στο κείμενο της έκθεσης. Παράγραφος 5, μετά το tense πρέπει να λέμε amounted αντί για amounts στα αγγλικά και γίνεται διαγραφή του φράσης as part of a global agreement ως μέρος ενός συνολικού ε, μια συνολική συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό στην παράγραφο 6. Αυτή είναι η διόρθωση και με αυτές τις προσαρμογές σας καλώ να εγκρίνετε την έκθεση με ονομαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ονομαστικά. Άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. 32 υπέρ και δύο Κατά. Δύο κατά, καμία εποχή. Και ευχαριστώ. Και μια τώρα μόνο ψηφοφορία σε σχέση πάλι με τη συνδιαλλαγή, το αποτέλεσμα συνδιαλλαγής, ειδοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2017 του Ζικφρίτ Μουρεσάν. και αυτή ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Καλώς, πέρας. Τριάντα υπέρ, δύο κατά δύο αποχές εγκρίνεται. Βάιντερε. Ταμείο Λεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία και μόνη ψηφοφορία και πάλι, ηλεκτρονικά και αρχίζουμε. Ψηφίσατε όλοι, πέρασε. Τριάντα δύο υπέρ. Δύο κατά. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Κυρία Βάιντερε. κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Από θεματικό, Είναι δική μου η πρόταση, πάλι, σε μία ψηφοφορία. Όχι, όχι. Με συγχωρείτε, σας τα μπέρδεψα, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν. τρεις τροπολογίες για την κινητοποίηση του ε, αποθεματικού έκτακτων αναγκών. Τροπολογία πρώτη, παράγραφος πρώτη, υπέρ. Τέσσερις. Κατά. Πολύ περισσότεροι αποχές απεριφθεί. Τροπολογία αριθμών 2, υπέρ. Τέσσερις πάλι, κατά. οι αποχές κανείς. Απερίφθη. Τρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Και πάλι. Αρχίζει. Πέρας. Τρεις ψήφοι υπέρ, τρεις, 30 υπέρ, τρεις κατά, μία εποχή. Και σας ευχαριστώ. Πόπα. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση επί από αίτηση της Φινλανδίας. Μια σειρά τροπολογιών υπαριθμών 2 έμπλ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία, πάλι της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα, Επιτροπή Απασχόλησης πάλι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. σε όρμα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έξι Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά ηλεκτρονικά καλύτερα αρχίζουμε μία ψήφος λείπει ακόμα Καλά, αν δεν θέλετε και να ψηφίσετε, δικαίωμά σας πέρα στις ψηφοφορίες. Απερίφθη. 14 υπέρ, 19 κατά, μία αποχή. Υπάρχει μόνο 7. Ε, Επιστροπή απασχόληση πάλι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται 8. Πάλι επιτροπή απασχόληση υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αριθμών 1 ζάορμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και λησμονήσαμε την έξι από ό,τι μου λένε Δεν ξέρω. Υπάρχει. Την ψηφίσαμε. Εντάξει, την καταψηφίσαμε. Δική μου ήταν η τροπολογία άλλωστε. Ναι, ναι, μην ανησυχείτε. Όλα υπό έλεγχο. Τελική ψηφοφορία της έκθεσης ε, ΠΟΠΑ ηλεκτρονικά. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται 31 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά. Και έχουμε και άλλο, άλλη μια ψηφοφορία για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση κατόπιν αιτήσω τη Ελλάδα αυτή τη φορά, Αττική συγκεκριμένα, με την κυρία Βιού. μια σειρά από τροπολογίε υπαριθμών. Δύο πρώτα απ' όλα Επιτροπή Απασχόληση υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτει η 3. Πάμε στην 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερη συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτει 1 τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά Πέρας. 31 ψηφί υπέρ, 3 ψήφοι κατά, εγκρίνεται και συγχαρητήρια. Και έκθεση Νόβακοφ. Εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Υπαριθμών 7, κόλμελ υπέρ. Κατά. Αποχές, απερίφθη. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία υπερθυμών ένα του εισηγητή Κύριε Νόβακο, τι θα μας πείτε. Μάλιστα, τίποτα. Αντιρρήσεις, όχι. Ψηφίζουμε το προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Α, θα ακολουθήσει η συμβαστική 1. Καλώ. Η 2 λοιπόν, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. απόχε. Εγκρίνεται. 10, 11, 12, 13 και 14 καταπίπτουν. Συμβαστική 3 υπέρ. Α, όχι, τη 13. Πρέπει να την ψηφίσουμε. Λάθος τα πω. 13 πρέπει να την ψηφίσουμε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 15, 16, 17 καταπίπτουν. Πάμε στη 18 του εισηγητή. Υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 20 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά ηλεκτρονικά καλύτερα αρχίζουμε πέρας απερίφθη 18 ψήφι κατά 15 υπέρ μία αποχή Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23, τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται ένα προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπαριθμών 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται φτάσαμε και στην συμβαστική υπαριθμόν. Ναι, υπέρ κατά Εγκρίθηκε η τρία έχει αποσυρθεί. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Καλώς. Μεταφορές. Θα δώσω το λόγο στον εαυτό μου. Αγαπητοί συνάδελφοι μου. 22, 27 και 31 μεταφορές. Θέλω να τις υποστηρίξετε. Την 28 την είχαμε μεταφέρει από την προηγούμενη συνεδρίαση. Είχαμε πει ότι δεν ήταν επαρκή η συνεργασία μεταξύ ΑΖΑ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευκρινίστηκαν το μεταξύ τα θέματα. Άρα προτείνω και την ε, μεταφορά 28. Να την υποστηρίξουμε. Στην 33 μόνο έχω μια ερώτηση για την Επιτροπή. Πρόκειται για προενταξιακή βοήθεια προς την Τουρκία που μας απασχόλησε πολύ στην ε, συνδιαλλαγή την Παρασκευή το βράδυ. Και αν θέλει να λάβει το λόγο η Επιτροπή για να μας εξηγήσει ο εκπρόσωπός της πώς προτείνεται μεταφορά κονδυλίων. Γιατί δεν το έχετε εντάξει μέσα στο αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής της Παρασκευής. Chair. Ευχαριστώ. Θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση αυτής της μεταφοράς ώστε να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για τα μέλη της Επιτροπής. Αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αίτηση μεταφοράς 62 εκατομμυρίων ευρώ στις πιστώσεις ε, ανάληψη υποχρεώσεων για το ενταξιακό μέσο για την Τουρκία ε, για ανθρωπιστική βοήθεια. Στις 16 Νοεμβρίου η Επιτροπή Προταξιακής ε, Βοήθειας ε, συνεδρίασε και έγκρινε τροπολογίες σε τέσσερα πολυετή προγράμματα για, το, ε, για τη συμφωνία με την Τουρκία. Και οι τροπολογίες αυτές αφορούν τη δημοσιονομική γραμμή από την οποία η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη οικονομική, κοινωνική και ταφική ανάπτυξη Τουρκίας χρηματοδοτείται. Δηλαδή Πρόκειται για την προενταξιακή γραμμή συνοχή για την Τουρκία, δημοσιονομική γραμμή. Λαμβάνονται υπόψη η έλλειψη ορίμαση κάποιων σχεδίων, καθώ και η έλλειψη στη... προβλήματα στη διαδικασία απορρόφηση, ιδιαίτερα στου τομεί όπω το περιβάλλον και οι μεταφορέ. Ω εκ τούτου και μετά τη συνεδρίαση τη σχετική επιτροπή, τα κονδύλια για το 2017 μειώθηκαν κατά 89 εκατομμύρια και οι υποχρεώσεις αυτές από τις 16 Νοεμβρίου ε, διατέθηκαν για την ε, ικανοποίηση εναλλακτικών αναγκών για το 2017. Η μείωση αυτή έγινε υπό το φως μιας ε, αποδεδειγμένης έλλειψης ικανότητας απορρόφησης εκταμίευσης για το 2017 και έγινε με τη σύμφωνη γνώμη των τουρκικών αρχών. Είναι σαφές λοιπόν ότι πρόκειται για ζήτημα δημοσιονομικής διαχείρισης αυτή η απόφαση της μείωσης ε, δεδομένης της αποδεδειγμένης ε, έλλειψης ε, της ικανότητας εκταμίευσης εκ μέρους της Τουρκίας. Ταυτόχρονα η ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία είναι ιδιαίτερως ανησυχητική και Πιστεύω ότι είστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την κατάσταση εκεί και τη γνωρίζετε. Ο αριθμό των εκτοπισμένων στη Συρία είναι 6,1 εκατομμύρια. 1,3 εκατομμύρια έχουν αφήσει τι αιστείε του πρόσφατα, ήδη τρέχοντο έτου του 2017. Και 13,5 εκατομμύρια εκτιμάται ο αριθμό των χρηζών των ανθρωπιστική βοήθεια. Για να ενισχύσουμε λοιπόν την ανθρωπιστική βοήθεια για την κρίση, προτείνουμε 62 εκατομμύρια από τα κονδύλια αυτά να αποδεσμευτούν από την ε, συμφωνία με την Τουρκία ε, στον ανθρωπιστικό προϋπολογισμό. Αν κατάλαβα σωστά την ερώτηση του κ. Γκάιερ, εδώ μιλούμε για το 2017, ενώ η συζήτηση της Παρασκευής αφορούσε τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, του 2018. Εν κατακλείδη, και για να σας προλάβω στην επόμενη σας συμπληρωματική ερώτηση, 89 εκατομμύρια απελευθερώθηκαν λόγω της μείωσης ε, του Γενικού Κονδυλίου της ΕΠΑ με την Τουρκία. Προτείνουμε λοιπόν μεταφορά 62 εκατομμύριων για την ανθρωπιστική βοήθεια. Οπότε η λογική ερώτηση είναι και το υπόλοιπο ποσό, τα 27 εκατομμύρια τι θα γίνουν. 17 εκατομμύρια από αυτά ενισχύουν ε, το ENI και ιδιαίτερα το μεσογειακό σκέλος, το νότιο σκέλος και αυτό που σας ενδιαφέρει είναι τα υπόλοιπα 10 ε, εκατομμύρια θα ενισχύσουν την UNRWA, τα Ηνωμένα Έθνη, ε, δηλαδή την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών που προσφέρει βοήθεια και αρρωγή στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Και μάλιστα Μερικέ μεταφορέ έγιναν εσωτερικά, δεν χρειάστηκε καν να υποβληθούν στην αρμόδια για τον προπολογισμό αρχή. Ε, ευχαριστώ. Τώρα εξηγούνται αρκετά. Γιατί το θέμα τη πρωταξιακής βοήθεια και η απόφαση που από τη συνδιαλλαγή ήταν μάλλον πολιτική αξιολόγηση. Ενώ εδώ μα λέτε ότι πρόκειται για μια απλή μεταφορά που έχει να κάνει με τη δυνατότητα απορρόφηση. Μπορώ να το δεχτώ, Απλώ. Στο 32 επίσης τη μεταφορά 32, σημαντικό ποσό, 77 και εκατομμύρια ευρώ. Πείτε μας λίγο ποιο είναι το υπόβαθρο, σας παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, το 10, 13, ε, 32, συγγνώμη, μεταφορά 32 αφορά ενίσχυση της, ε, του τοπικού μέσου για την ενέργεια το, του μέσου Ελένα, όπως προβλέπουν τα αρχικά, που το διχειριζόμαστε δυνάμει του ορίζοντας 2020. Προτείνουμε 77,3 ε, εκατομμύρια μεταφερθούν από το ενεργειακό σκέλος του συνδέοντος στην Ευρώπη για να ενισχυθεί αυτό το μέσο Ελένα. Η ενίσχυση του Ελένα είναι μια συνέχεια της ανακοίνωσης ε, της καθαρής ενέργειας για όλους τους Ευρωπαίους της 30 ε, Νοεμβρίου του 2016. Και θέλουμε να απελευθερώσουμε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον κατασκευαστικό κλάδο. Επίσης, η ενίσχυση αυτού του, της ευρωπαϊκής υποστήριξης τοπικής ενέργειας από ε, τα, ε, από τα κονδύλια αυτά μέσω του ορίζοντα προ, προτείνεται σε δύο δόσεις. 77 εκατομμύρια για το 2017 και για το 2018 επίσης θα έχουμε μια μεταφορά της αρμόδιας για το προπολογισμό αρχής, αλλά την περασμένη Παρασκευή ήδη το προλάβαμε ε, συμπεριλαμβάνοντας το αμέσως στα συμπεράσματα ε, της Επιτροπής Ιδιαλλαγής. Δηλαδή αυτά τα 20 εκατομμύρια ήδη περιλαμβάνονται στον, προτα... προπολογισμό ως ε, μείωση του... της ασφαλούς ενέργειας και του ορίζοντας 2020. Ευχαριστώ πολύ. Ρίχνω μια, μια ματιά στους συναδέλφους αν θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε. Κάποια διευκρίνηση όχι. Καλώς. Ως εισηγητής λοιπόν προτείνω την έγκριση όλων των μεταφορών. Και η γραμματεία μου λέει ότι μπορούμε και ε, ομού να τις ψηφίσουμε μεν ηλεκτρονικά δε, εάν δεν έχετε αντιρρήσεις. Όχι. Αρχίζουμε την ψηφοφορία λοιπόν για τις μεταφορές. Πέρας. 26. μία ψήφο κατά δύο αποχές και σας ευχαριστώ πολύ. Και περνούμε στα ε, άλλους, στα άλλα τμήματα με τον κύριο Τάραντ. Κύριε Τάραντ, ε, να μας πείτε αναθεσμικό όργανο τι προτείνετε. Γιατί βλέπω ότι δεν είστε διατεθειμένος να υποστηρίξετε κάποιες μεταφορές και θα είναι καλύτερο και πιο διαφανές για μας να έχουμε μια εικόνα ανά όργανο. Παρακαλώ, αναθεσμικό όργανο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα το κάνω όπως ακριβώς προτείνεται. Αλλά με μια μικρή αλλαγή. Πρώτον, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άκουσα ότι η στρατηγική της Επιτροπής να μειώσει το κόστος των κτηρίων στην συνδιαλλαγή έγινε, λέγω, βλέπω επιπτώσεις αρνητικές και στο δικαστήριο και ακόμα και αν έχουμε τις ευλογίες της κυρίας Χολμάιερ θα ζητούσα από τους συναδέρφους να επιτρέψουν τη μεταφορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ιδιαίτερα τη μεταφορά για τα κτίρια. Και αν σας κατάλαβα καλά, Πρόεδρε, πρώτα θα ψηφίσουμε ή θέλετε να περάσω στα υπόλοιπα και να μιλήσω και για τα άλλα θεσμικά όργανα. Ναι, ναι, να μιλήσετε Προτιμώ ένα θεσμικό όργανο, Τότε μπορούμε να ψηφίσουμε για το δικαστήριο τώρα και μετά να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, εφόσον επιθυμείτε βεβαίως ακολουθείτε και την πρόταση του εισηγητή. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ψηφίζουμε. Το τέλος, οπότε σε ακούμε για τα υπόλοιπα. Ωραία. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είπαμε, και έχουμε και τέσσερις μεταφορές, τρεις από τις οποίες είναι συνήθεις μεταφορές. Υπάρχει 14 και θέλω να επιστήσω την προσοχή των συναδέρφων εδώ στο γεγονό ότι λυπούμε αλλά δεν μπορώ να το στηρίξω γιατί λέει ότι το περισσότερο προσωπικό στο Λουξεμβούργο υποφέρει από προβλήματα πλάτης, μέσης και γι' αυτό χρειάζονται ηλεκτρικού τύπου γραφεία. Ε, τι να πω, πάντα στηρίζω την δημιουργία καλύτερων συνθήκων εργασίας για τους ανθρώπους που κάνουν σκληρή δουλειά αλλά μετά μάθαμε ότι 716,10 ευρώ στοιχίζει κάθε τέτοια ηλεκτρική καρέκλα, μα τόσο πληρώνεται στην Εστονία ένας δάσκαλος. Ξέρω ότι το Λουξεμβούργο είναι μια ακριβή χώρα, αλλά ίσως θα ήταν προτιμότερο, τι να πω, ας ε, νοικιάσουμε καλύτερα κάποιον γυμναστή, κάποιον ε, για να βοηθήσω του ανθρώπου αυτού. Έχουμε εμεί εδώ ηλεκτρική. Και εμένα, εγώ υποφέρω από τη σποδηλική μου στήλη. Έχω εγώ ηλεκτρική καρέκλα. Οπότε καλύτερα να τα δώσω στο Κλάου Βέλε τα χρήματα αυτά για να κάνει κάτι για του ευρωβουλευτέ. Αντί για το προσωπικό του ελεγκτικού συνεδρίου που έχει προβλήματα με την πλάτη του. Και εδώ δεν το λέω με ηρωνία. Προσέξτε. Σε πόσο μακριά θα πάμε. 716 το καθένα. Το φαντάζεστε ο κόσμος στο Λουξεμβούργο ίσως θα έπρεπε να κάτσει να ξανασκεφτεί τι ζητάει. Άλλοι υποφέρουν περισσότερο. Και αυτοί χρειάζονται ηλεκτρικά, ηλεκτρικό εξοπλισμό. Μπορεί να μην είμαι πολιτικά ορθός και ζητώ εκ των προτέρων ε, συγγνώμη, αλλά αν είναι έτσι, τότε να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρική καρέκλα όπως χρησιμοποιούν στις Ηνωμένε Πολιτείες. Τι να πω. Αφού δεν το εννοείς ηρωνικά, το γράφουμε και στα πρακτικά. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που είπες. Με την αυτή διαδικασία. Συμφωνείτε. Ψηφίζουμε. Η πρόταση είναι τρεις μεταφορές του ελεγκτικού συνεδρίου να γίνουν δεκτές, η 14 να απορριφθεί. Αυτή είναι η πρώτη του εισηγητή σα. Λοιπόν, το πάμε σιγά σιγά. Πώς, ποιος είναι υπέρ της θέσεως του εισηγητή υπέρ της έγκρισης αυτών. Η 14 απορρίπτεται από τον εισηγητή για το ελεγκτικό συνέδριο. Αυτή θέλει να απορρίψει ο Ίντρεκ. Προτείνω λοιπόν την 11, 12 και 13 να τις ψηφίζουμε ομού. Τις υποστηρίζω εισηγητής. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Χωσέ Εμμανουέλ. Για, να τα καταλάβουμε κάπως καλύτερα. Δεν είναι πιο εύκολο να ψηφίσουμε μόνο τη μεταφορά 14. Και αν ψηφίσουμε ναι, ψηφίζουμε υπέρ της μεταφοράς. Αν ψηφίσουμε όχι, αυτό προτείνει ο συγκητής δηλαδή. Αν ψηφίσουμε ναι, να ψηφίσουμε να εγκρίνουμε τη μεταφορά, αλλιώ όχι, ουσιαστικά είμαστε με τη θέση του εισηγητού. Είναι πιο απλή έτσι νομίζω η διαδικασία. Dann κύριο Γκάιερ. Καλώ. Ακολουθούμε τότε την πρόταση του Χωσέ Μανουέλ. Μου φαίνεται πολύ λογική. Έτσι, για να είμαστε σίγουροι τώρα ότι συνοηθήκαμε. Δεν υπάρχει αντίρρηση ω προς την 11-12-13, εντάξει. Ωραία. ωραια Επομένω, τώρα ψηφίζουμε την μεταφορά υπαριθμών 14, για την οποία ο εισηγητή σα προτείνει να απορριφθεί. όποιο πει ναι, ακολουθεί την κύριο Τάραντ, λέει ο μιλητή. Όποιο όχι, αντιτίθεται στην πρόταση του κυρίου Τάραντ. Ένα λεπτό, εδώ έχουμε ένα, ένα αίτημα, έτσι, μια πρόταση. Εδώ είναι ο συγητής. Η δική του η τροπολογία είναι απορρίπτουμε αυτήν την μεταφορά. Όποιο τον υποστηρίζει ψηφίζει το πράσινο. Όποιο δεν τον υποστηρίζει πατάει το κόκκινο. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, να μην τα μπερδέψουμε πολύ στη διαδικασία, το κάνουμε ανάποδα, το πιάσουμε παλιό. Η Επιτροπή δέχεται την απόρριψη αυτού του αιτήματος μεταφοράς. Μα αυτό σας λέω. Πρέπει να ψηφίσουμε την πρόταση του εισηγητή. Λοιπόν, αντιελεκτρονικά. Ίντρεκ. Ο Ίντρεκ προτείνει να απορριφθεί η μεταφορά. Ο Ίντρεκ προτείνει την απόρριψη της μεταφοράς. Δηλαδή, εσείς ΕΛΚ που λέτε όχι, θέλετε να, να εγκριθεί η μεταφορά, έτσι. Εγκρίνεται η μεταφορά, έτσι. Για να είμαστε σίγουροι ότι καταλάβαμε. Καλώς, ομόφωνα λοιπόν ε, εγκρίνεται και απορρίπτεται εν το άμα. Καλά, εντάξει, προχωρούμε, δικό μου το λάθος. Attends, euh, on va mettre... C'est Κύριο Σκάιερ, λοιπόν, εάν καταλαβαίνω καλά, με το ότι καταψηφίσατε τον Ίντρεκ, εγκρίνατε τη μεταφορά. Ωραία. Και έτσι πάμε στο τελευταίο θεσμικό όργανο. Ο κύριος Δενανό, πρόεδρε, είναι... Πράγματα είναι πιο απλά. Θα πρέπει να πούμε υπέρ ή κατά της μεταφοράς. Αν είμαστε υπέρ της μεταφοράς ψηφίζουμε υπέρ, αν είμαστε κατά της μεταφοράς ψηφίζουμε κατά. Also. Ich bin ja eurer Ansicht, nur kriege ich von hier... Και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αλλά η γραμματεία μου τα λέει αλλιώς. Για να μας τα εξηγήσετε λοιπόν εσείς. José Manuel, Bon. Ή μάλλον ο Χωσέ Μανουέλ. Καλά, ας Δεχτούμε την πρόταση του Πρόεδρου. Δέχομαι την πρόταση του Πρόεδρου. Ο Πρόεδρος δεν θα θέσει σε ψηφοφορία τη μεταφορά καθ' αυτή, αλλά την πρόταση του εισηγητού, του κυρίου Τάραντ. Επί της προτάσεως Τάραντ θα ψηφίσουμε, που είναι και ο εισηγητής. Αυτό πρότεινε ο Πρόεδρος. Οπότε εμείς θα ψηφίσουμε, που είμαστε υπέρ της μεταφοράς, θα ψηφίσουμε κατά της πρότασης του εισηγητού. Αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ψηφίζουμε αν ψηφίσετε υπέρ της πρότασης του εισηγητού, είστε κατά της μεταφοράς. Εμείς όμως είμαστε υπέρ της μεταφοράς, άρα θα ψηφίσουμε κατά της πρότασης του εισηγητού. Τα πράγματα είναι φως φανάρι. Okay, also, das war mein Vorschlag von vor ungefähr 10 Minuten. Πριν από 10 λεπτά πάλι εγώ αυτό σας είχα πει, το ίδιο είχα πει ακριβώς και ευχαριστώ για τη διευκρίνηση, λέει ο Πρόεδρος. Να τα πω στα αγγλικά, πως με καταλάβετε καλύτερα. Μόιντρεκ προτείνει όχι για την μεταφορά αριθμός 14. Ηλεκτρονικά λοιπόν θέτουμε το ερώτημα ποιος στηρίζει τον εισηγητή. Εντάξει. Όποιος δεν θέλει να στηρίξει την πρόταση του εισηγητή πρέπει να ψηφίσει κατά. Εντάξει τώρα, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Τελείως, αυτό θα κάνουμε.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 ψήφι κατά. Απερίφθη, άρα επικυρώνεται η μεταφορά. Indrex lost. Yeah, they get the electronic. Ωραία, θα τους δώσουμε τις ηλεκτρονικές, ηλεκτρικές, πώς τις θέλετε αυτές οι καρέκλες. Α, γραφεία, καλά. Εντάξει, Indrek, τελειώσαμε. Όχι, προχωράς. Αγαπητοί συναδελφοί, συγγνώμη που δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Τι να πω, εγώ έτσι καταλαβαίνω τα περί μουσικών καρεκλών. Α, ηλεκτρικών, συγγνώμη, διορθώνω, λέει ο κύριο Τάραντ. Τώρα λοιπόν συνεχίζουμε και περνάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι πάντα πολύ σημαντικό. Διότι Ευτυχώς έχουμε και τον κύριο Κλέτη εδώ, που θα μπορούσε ίσως να απαντήσει σε δύο ερωτήσεις που έχω. Απορρέουν από το γεγονός ότι στην Επιτροπή Προπολογισμών δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να ανταλλάξουμε πληροφορίες όπως θα θέλαμε. Πρώτον λοιπόν, μπορούν να μου πούνε οι υπηρεσίες κατά πόσο υπάρχει άλλη δυνατότητα χρηματοδότηση των μεταφορών 3 και 4 και όχι από τα κτίρια, από τους τρεις χώρους εργασίας. Γιατί δεν θα ήθελα να έχουμε πάνω από 7 εκατομμύρια να τα αφήσω στην τύχη μελλοντικών μεταφορών. Ο κύριος Σάσουετ. τα βρίσκουμε καλά. Εντάξει, εγώ δεν το βάζω σε εσά γιατί δεν θέλω να βάλω σε εσά το βάρος να απαντήσετε. Τέλο πάντων και το άλλο. Γιατί τα σχέδια εξοπλισμού δεν συμπεριλήφθηκαν στο φετινό προπολογισμό. Λέτε ότι θέλετε να αφήσετε το προπολογισμό σε αποδεκτά επίπεδα. Και αυτό θα έπρεπε να είναι πάντα οι πραγματικές ανάγκες για τον προπολογισμό ή κάνω λάθος. Λοιπόν, αυτά τα δύο θέλω να ρωτήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι κανείς εδώ από τη διοίκηση που μπορεί να δώσει απαντήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σας δώσω τις σωστές απαντήσεις. Λοιπόν, ρωτάτε αν μπορούμε να ε, κάνουμε τη μεταφορά τρία και τέσσερα από άλλες γραμμές. Θεωρητικά ναι, αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα, μια δυσκολία που θα έχει σαν αποτέλεσμα ότι αν έρθει σε εσά στις 4 Δεκεμβρίου τότε θα έχουμε προβλήματα και μετάφρασης και διερμηνίας προκειμένου να παρουσιάσουμε μια άλλη πηγή. Και θα εξηγήσω γιατί ισχύει αυτό για το σε 3 και το σε 4. Γιατί δηλαδή τα 7 εκατομμύρια θα ήταν καλύτερα να τα πάρουμε από τη διευθέτηση χώρων. Είναι μια γραμμή η οποία αρχικά είχε 84,5 εκατομμύρια και κινητοποιούμε 9% της γραμμής αυτής που εκτιμήθηκε το Δεκέμβριο του 2015 για την αίσθηση του 2017 και τώρα είμαστε στο τέλος του 2017. Υπάρχει λοιπόν το θέμα του χρόνου. Όταν στα τέλη του 2015 καθορίζουμε τον προπολογισμό για τους τρεις χώρους εργασίας και για το σύνολο των γραφείων πληροφοριών στις διάφορες πρωτεύουσες, υπάρχει αβεβαιότητα για κάποια σχέδια που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Και υπάρχει και ένα δεύτερο γενικό πρόβλημα που θα ήθελα εδώ να αναφέρω και που είναι η σημαντική προσπάθεια που έγινε στον τομέα των ε, έργων που σχετίζονται με την ασφάλεια. Βλέπετε το 2017 τι έγινε στο Στρασβούργο κυρίως. Συνεπώς κινητοποιούνται οι ομάδες για αυτά τα κατά έργα που εσείς αναγνωρίσατε ως τέτοια προτεραιότητας όταν ε, καθορίσατε τον προπολογισμό των δύο τελευταίων ετών. Αυτό σημαίνει επίσης ότι κάποια στιγμή ε, σχέδια μικρότερης προτεραιότητας δεν έχουν αρκετό προσωπικό για να υλοποιηθούν. Και θα σας πω ποια είναι αυτά ή ποιε είναι οι συνθήκες που έχουν σαν αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε 7 εκατομμύρια για αυτή τη γραμμή διαθέτησης χώρων. Κυρίως στις Βρυξέλλες. Το πρώτο σύνολο σχεδίων έχει να κάνει με την έλλειψη απόφασης για το κτίριο PHS. Εκεί γίνονται προπαρασκευαστικές εργασίες που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά της βιβλιοθήκης και του γραφείου του Πρόεδρου και του Γενικού Γραμματέα αλλά και άλλων υποδομών. Και επειδή δεν ελήφθη απόφαση για το PHS, αυτές οι προκαταρτικές εργασίες, μελέτες κτλ. δεν έχουν ε, ξεκινήσει. Στη συνέχεια, εκτάκτος, είχαμε ένα έσοδο για το Square Mails με σύμβαση. Δηλαδή έγιναν τα έργα και όταν ε, παίρναμε το κτίριο έπρεπε να μας επιστρέψει ο εργολάβος 2 εκατομμύρια, άρα έχουμε φτάσει στα 3. Επίσης έχουμε και μια καθυστέρηση στην, ε, στο για προσφορές για τις Βρυξέλλες γενικά όσον αφορά την πυρασφάλεια. Αυτό δεν είναι τόσο σοβαρό, αλλά σε ένα διαγωνισμό δεν πετυχαίνετε πάντα το χρονοδιάγραμμα όπως θέλετε γιατί δεν το χειρίζεστε εσεί. Επίσης για μια αίθουσα σεμιναρίων στο Άτριουμ καθυστέρησε που είναι 800.000 ευρώ. Επίσης αναβλήθηκαν ε, σχέδια έργων στο κτίριο Τρεβ γιατί ανάμεσα στα τέλη του 2015 και τώρα αποφασίστηκε να γίνει ανακαίνιση του συνόλου του κτηρίου Τρέβα το 2020, οπότε είναι περιττό να ξεκινήσουν τώρα να γίνονται κάποια επιμέρους έργα. Αυτά όσον αφορά τα κύρια έργα στις Βρυξέλλες. Ήδη έχουμε φτάσει εδώ στα 5,5 εκατομμύρια. Στο Λουξεμβούργο από την άλλη μεριά. Εγκαταλείψαμε κάποια μικρά έργα γιατί η προοπτική μετακόμισή του ΚΑΝΤ πλησιάζει. Οπότε δεν έχει νόημα. Μπορεί να υπάρξουν ε, διαιτησίες και για το Σούμαν. Στο Στρασβούργο επίσης υπάρχουν ε, διάφορα έργα διευθέτηση που καθυστέρησαν, γιατί οι ομάδες αφοσιώθηκαν πλήρως στα μεγαλύτερα έργα ασφάλειας όσον αφορά την είσοδο του κτηρίου WIC. Βλέπετε πόσο προχωράνε τα έργα. Και η τελευταία θέση που μας εξασφαλίζει πόρους είναι το Γραφείο Πληροφοριών στο Παρίσι. Είχαμε προβλέψει 2 εκατομμύρια όταν θέτασε στη διάθεση του Κοινοβουλίου το γραφείο αυτό, αλλά στις τελικές διαπραγματεύσεις για το σχετικό συμβόλαιο προβλέπεται και ε, επιστροφή. 2 εκατομμύρια παραπάνω λοιπόν προβλέπονται εδώ. Τέλος, φτάνουμε εύκολα στα 7 εκατομμύρια που είναι στην ε, διάθεσή μας για τη μεταφορά αυτή, για την μεταφορά επίσης των υπολείπων προς εκαθάριση που θα σας παρουσιάσουμε στις 4 Δεκεμβρίου στην τελευταία σας συνεδρίαση. Δεν υπάρχει λόγος να αρνηθούμε κονδύλια για μία γραμμή και να επιμείνουμε να τα αφήσουμε σε μία άλλη. Τέλος για τις επενδύσεις που είναι το 4 και το 5 στην πραγματικότητα. 5 και 6 Στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό προσπαθούμε να περιορίσουμε την αύξηση του προϋπολογισμού και είμαστε στο 1,7-1,8% τα τελευταία χρόνια όσο και ο πληθωρισμός. Βέβαια υπάρχουν ε, σχέδια επενδύσεων γνωστά, αλλά είναι δύσκολο να τα προσθέσουμε αν θέλουμε να μείνουμε στα επίπεδα του προπολογισμού του περιορισμένου όπως μας έχει υποβληθεί. Με τα 2 δισεκατομμύρια έχουμε ένα πλεόνασμα τεχνικής φύσεως στα τέλη της χρονιάς της τάξης του 2%. Οπότε η ιδέα είναι να ολοκληρωθούν οι δημοσιονομικές συζητήσεις επί του προϋπολογισμού με στόχο την άνοιξη, ξέροντας ότι αν υπάρξουν απαραίτητα ανάγκε επενδυτικές γίνεται με την άδεια της αρχής επί του προπολογισμού και γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα μπροστά σας, μπορούν να γίνουν με τα πλονάσματα στα τέλη της χρονιάς. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να παραμείνουμε στα όρια του προπολογισμού, αλλά να αποφεληθούμε και από μια ευελιξία περιορισμένη στο 10% του προπολογισμού. Και εδώ για τις επενδύσεις θα έλεγα είμαστε κάτω από 1% του ετήσιου προπολογισμού. Οπότε ο δημοσιονομικός κανονισμός την προβλέπει την ευελιξία αυτή και άρα υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς πιστώσεων εφόσον την εγκρίνει η αρχή επί του προπολογισμού. Ευχαριστώ. Μας κάνει και τη σύσταση ο εισηγητής. Σας ευχαριστούμε κύριε Κλέτη. Μάξιμα σουφίτσιτα, όπως θα έλεγε και ο καθηγητής μου. Είμαστε υπέρ. Okay. Άρα δέχεται, υποστηρίζει μάλλον αυτή την μεταφορά, δεν βλέπω αντιρρήσει, εγκρίνεται και συγχαρητήρια. Και κτίρια, κτίρια Συγγνώμη, συγγνώμη, θα ήθελα να προσθέσω κάτι ως πρόταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών ε, οι εισηγητές του επόμενου έτους θα είναι ο κύριος Άσχορθ, εγώ και ο περσινός ε, εισηγητής για τις μεταφορές. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η συνεργασία ε, στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης του προϋπολογισμού. Να γίνει δηλαδή ένας ενδελεχής έλεγχος των προτάσεων των θεσμικών οργάνων. Γιατί ε, οι μεταφορές ε, δείχνουν εξορισμού ότι μερικές δημοσιονομικές γραμμές είναι υπερεπαρκής και εσκεμένα έχουν ε, προγραμματιστεί ποσά για την για τον αρτασμό της επαιτίου του ελεκτικού συνεδρίου και το καθεξής. Οπότε είναι σημαντικό ο εισηγητής ε, του επόμενου έτους να γνωρίζει αυτές τις πληροφορίες, τις διαπραγματεύσεις που θα έχει με τα θεσμικά όργανα του χρόνου. Καλώς, κτηριακή πολιτική. Αλλά από ό,τι μου λένε δεν πάμε στην... Όχι, δεν είναι η Μαρίζα. Οπότε, εντάξει. Διάφορα. δεν υπάρχουν. Και υπενθυμίζω ότι αύριο αρχίζουμε 8 και 30. Έτσι, ευχαριστώ και πέρα συνεδρίασης.